Sí, buenas tardes a todos. Pido que vayan tomando. Καλό σα απόγευμα. Παρακαλώ να καθίσετε στι θέσει σα γιατί θα ξεκινήσουμε με τη συνεδρίασή μα. Bueno, buenas tardes. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους και πάλι. Παρακαλώ λίγη ησυχία αν γίνεται. En primer lugar, tenemos el Πρώτα απ' όλα έχουμε το σημείο 1 στην ημερήσια διάταξη, που είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Και αν δεν υπάρχουν τροποποιήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη ως έχει. Μετά, σημείο 2. Η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 22 <clears throat> και 23 Νοεμβρίου. Αν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης ε, δεν θα υπάρξουν παρατηρήσεις, ε, θα εγκριθούν αυτά τα πρακτικά, θα θεωρηθεί ότι κυρώνονται. Στη συνέχεια έχουμε το σημείο 3, ανακοινώσεις της Προέδρου. Και θα ήθελα να σας ανακοινώσω σε όλους ότι η κυρία Αντρές Μπαρέα της Σοσιαλιστικής Ομάδας έπαψε να είναι μέλος της Επιτροπής Αλληλείας στις 15 Δεκεμβρίου και πέρασε στην Επιτροπή Ενέργειας, Έρευνας, και αντικαθίσταται την κυρία Ντολόρες Γκαρσία Γέρο Καραβάγιο, πάλι επίσης από την Σοσιαλιστική Ομάδα, που είναι μία από τις καινούργιε ευρωβουλευτίνες που ήρθαν τώρα ως παρατηρητές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα εξ ονόμας να καλωσορίσω την, να χαιρετήσω την κυρία Ανδρές Μπαρέα και να την ευχαριστήσω για συνεργασία και να καλωσορίσω την αντικαταστατριά της και στην κυρία Ανδρές Μπαρέα εύχομαι κάθε επιτυχία. Ήταν είναι ο τελευταίος αποχαιρετισμός του κοκτέιλ και καλωσορίζουμε την κυρία που την αντικαθιστά και ελπίζουμε ότι θα είναι Είμαστε βέβαιοι θα είναι τόσο καλή και συνεργάσιμη όπω ήταν η κυρία Αντρε Μπαρέα. Λοιπόν, με αυτά περνάμε στο σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη, που είναι το πρωτόκολλο που συμφωνήθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία τη Γουινέρ Μπισάου που καθορίζει τις αλληλευτικές δυνατότητες και την χρηματική αντιπαροχή και αντιστάθμιση που προβλέπεται από την αλληλευτική σύμπραξη. Εισηγητής ο κύριος Χόγλοντ. Πρόκειται πάλι για μια παράταση του πρωτοκόλου Κύριε Χάγκλοντ, έχετε τον λόγο λοιπόν τώρα. Ή όχι, καλύτερα. Έχετε εσείς τον λόγο κύριε Χάγκλοντ λοιπόν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως περιγράφηκε από την πρόεδρο, έχουμε μία παράταση ενός έτους αυτού του πρωτοκόλου που θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο 2012 και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πάλι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου βρισκόμαστε πίσω σε σχέση με τα θέματα αυτά και πρέπει να μπορεί το Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί εκ των υστέρων αντί ε, εκ και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε στο μέλλον για να αποφύγουμε δυσκολίες και δυσχέρειες σε σχέση με τέτοιου είδους πρωτόκολλα. Αλλά αυτού του είδους είναι η πιο κριτική παρατήρηση. Έχω όμως και πιο θετικές παρατηρήσεις. Η συμφωνία αυτή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 και ε, η αναλογία ε, είναι θετική σε σχέση με τα αποθέματα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται να έχουμε μια σχετικά σταθερή κατάσταση όσον αφορά τα τα αποθέματα αλλιευμάτων. Καλό πράγμα αυτό, προϋπόθεση για να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία. Και βλέποντας την έκθεση αξιολόγησης, ωστόσο, από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποια προβλήματα με κάποια στοιχεία. Είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε ότι η ποιότητα αυτών των στοιχείων κτλ. θα βελτιωθεί στο μέλλον για να διασφαλίσουμε έτσι ότι τα συμπεράσματα που θα συνάγονται όσον αφορά τα αποθέματα θα είναι ικανοποιητικά και θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το κέρδος ε, σε σχέση με την απασχόληση μετριοπαθές ε, έχουμε το συμπέρασμα ότι μια και η Γουινέα Μπισάου είναι μια από τις φτωχότερες χώρες παγκόσμια θα μπορέσει να υποφεληθεί. Έχουμε και την, το, Ταμείο της Ευρω... το Ταμείο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η συμφωνία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για αυτή τη χώρα οικονομικά. Η συμφωνία για την Αλία είναι 7,3% των συνολικών κυβερνητικών εσόδων για την Γινέα Μπισάου και 88% όσον αφορά την αλληλεία. Και είναι σημαντικό να έχει αυτή τη συμφωνία αυτή η χώρα. Γενικά λοιπόν αυτή είναι η συμφωνία. Ελπίζω να έχετε εξοικειωθεί με τη σύντομη εισαγωγή μου με αυτήν. Η σύστασή μου είναι το Ευρωκοινοβούλιο να εγκρίνει, να συνενέσει με την παράταση του πρωτοκόλου και ελπίζουμε φυσικά στη συνέχεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει από πλευρά τη μια πιο μια ευρύτερη από πλευράς χρονικής διάρκειας συμφωνία και σε σχέση με την υποβολή της θα πρέπει έγκαιρα να υποβληθεί, να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο, ώστε να έχουμε τον χρόνο να την εξετάσουμε, να την δούμε, προτού αρχίσει να ισχύει, υποθέτω, του χρόνου. Αυτά είχα να πω, κυρία Πρόεδρε. Θα έπρεπε να συνενέσουμε, να εγκρίνουμε και δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τους ε, βοηθούς και την γραμματεία και τα μέλη της διοίκησης για τη βοήθεια που μου παρέσχουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Lundgren, Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ήταν εξαιρετική αυτή η εισαγωγή, αυτή και για την απόφαση του Συμβουλίου που έχω εδώ μπροστά μου στα αγγλικά Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Χόγκλουντ ότι αυτή η συμφωνία είναι πραγματικά βελτιώνεται, μπορεί να βελτιωθεί. Uh, η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ρήτρα για το πάγωμα την κατάλληλη την άρση αυτής της συμφωνίας σε περίπτωση παραβιάσεων είναι αυτό που πρέπει να προσπαθούμε να πετύχουμε. Είναι μια συμφωνία που παρέχει εισόδημα και είναι πολύ σημαντική για αυτόν τον λόγο για την Γινέα Μπισάο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι υπεύθυνη, με υπεύθυνο τρόπο να προσεγγίσει τις ευκαιρίες που έχει να αλλιεύει στα ύδατα, χωρικά ύδατα της χώρας αυτής, της Γουινέας Μπισάο. Έχω κάποιες ερωτήσεις για την ίδια τη συμφωνία και θα ήθελα να ξεκινήσω ε, στρεφόμενοι προς το άρθρο 5 που προβλέπει την αναθεώρηση των αλλιευτικών δυνατοτήτων. Αν η Επιστημονική Επιτροπή που θα πρέπει να συνέρχεται κάθε χρόνο θεωρήσει ότι μπορεί να υπάρχει κάποια, κάποιος χώρος για αύξηση των δυνατοτήτων αλίευσης, η χρηματοοικονομική συνεισφορά που πληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και αυτή να αναλογικά να αυξηθεί. Και όταν πρόκειται για το διπλάσιο κατά μέγιστον όπως στο άρθρο 2 αντί για 4 εκατομμύρια έχουμε, θα έχουμε και το 14 εκατομμύρια διπλάσιο δηλαδή ε, όγκο αλλιευμάτων που α, αφορούν αυτή τη δυνατότητα. Η ερώτησή μου είναι από ποιο ταμείο θα βρούμε τα πρόσθετα κονδύλια έχουμε περιορισμένα κονδύλια για τέτοιου είδους συμφωνίες αλληλείας. Ίσως μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει κάπως καλύτερα τι συμβαίνει σε σχέση με αυτό το άρθρο. Και για το άρθρο 6 στη συνέχεια, 6 εδάφιο 5. 6 εδάφιο 5. Ναι. Κάνει λόγο για δυνατότητες διακρύβωσης διερευνητικά αλληλευτικών δυνατοτήτων και στο 5 λέγεται τα αλλιεύματα κατά τέτοιου είδους ε, διερευνητικές δυνατότητες θα πρέπει να είναι υποκυριότητα των ιδιοκτητών του σκάφους ε, και σε σχέση με ε, τέτοιου είδους αλλιεύματα που δεν επιτρέπονται να αλλιεύονται ή να τίθενται σε εμπορία Διερωτώ με πώς μπορούν να αποφύγουν τέτοιου είδους αλλιεύματα αυτά τα σκάφη που απαγορεύονται υπό την νομοθεσία της Γουινέας Μπισάου. Πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η συγκεκριμένη πρόκληση. Και ένα άλλο άρθρο, το οποίο με το θεωρώ αξιοπερίεργο, είναι το 7α για ασυνήθιστες έκτακτες συνθήκες ε, όσον αφορά τις αλλιευτικές δραστηριότητες ε, που θα παρακόλλιαν ε, αυτές και ότι τότε θα έπρεπε ίσως να μην πληρώνονται αυτές οι αντισταθμίσεις. Ποιες θα ήταν αυτές οι έκτακτες προϋποθέσεις εκτός από θεομηνίες ή φυσικά τέτοια μετεωρολογικά φαινόμενα κτλ. Πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη ρήτρα αυτή που αναφέραμε, τι θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Έχετε κάτι υπόψη από πράσινη επιτροπή, πειρατεία για παράδειγμα, τι θα μπορούσε να ήταν αυτό. Νομίζω λοιπόν ουσιαστικά με αυτές τις παρατηρήσεις καλύπτομαι. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω εξ ονόματος της Επιτροπής ο κύριος Βέρκε θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε βουλευτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε τον για την παρουσίαση της εκθεσής του. Πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντική η συζήτηση και η συζήτηση που έχουμε σήμερα όσον αφορά το πρωτόκολλο αυτό για την αλληλεία. Αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να κάνω αυτή τη στιγμή μια διευκρίνηση όσον αφορά τα ίδια εκείνα τα οποία άπτονται αυτή τη συνθήκη δεν έχουμε τα πελαγικά ψάρι, ψάρια, αλλά περισσότερο είναι, η αξία η μεγαλύτερη είναι σε σχέση με τα κεφαλόποδα και τα οστρακοειδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή οστόλο και τη δυνατότητα λίευσης, οι οποία προβλέπεται για τον το Θα σας δώσω τόνει, Θα σας δώσω τους αριθμούς, γνωρίζετε βεβαίω από αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα μεικτέ αυτές συμφωνίες που γίνονται έρχονται σαν ένα παράρτημα όσον αφορά τις πρωτο, πρωτοβουλίες οποίες, και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί. Υπενθυμίζω ακόμη πως ε, ότι έχουμε 4.400 για τις 4.400 τεζιμπέ για τα κεφαλό ποτά καθώς επίσης το ίδιο ποσό όσον αφορά τις γαρίδες. Επίσης, επίσης άλλα τόσα όσον αφορά τα ύδατα της γυνές Γουινέας Μπισάου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα βασικά της συμφωνίας αυτής. Το υπογραμμίσατε. Τα στοιχεία και τα επιστημονικά τα οποία έχουμε χείρε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε εμεί να σταθεροποιήσουμε του πόρου αυτού του αλληλευτικού οι οποίοι μα ε, βοηθούν πολύ για να προσπαθήσουμε να θέσουμε λειτουργία ενισχύει αυτή τη συμφωνία και η σχέση που έχουμε με τη χώρα αυτή για την ανανέωση της συμφωνίας αυτής και να υπάρξει μια διάσταση επιστημονική και αυτή η διάσταση να εγγραφεί πεντακάθαρα καθώς επίσης και δραστηριότητες μιας κοινή επιτροπή η οποία θα ασχολείται με τα πανεπιστημονικά θέματα. Ποια θα είναι η δράση της, ποια η δραστηριότητά της, ποια ο ρόλος της. Αναφερθήκατε επίσης, μεταξύ άλλων, στη νέα ρήτρα όσον αφορά το προηγούμενο συνθήκη που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το οποίο βεβαίω έδινε τη δυνατότητα αναστολή αυτή τη συμφωνία εφόσον υπήρξε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών. Όντω, αυτή είναι η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κομισιόν για να υπάρχει πάντοτε αυτή η ρήτρα στο σύνολο των συμφωνιών οι οποίε γίνονται στον τομέα τη αλληλεία και επιμείναμε εμεί να υπάρξει αυτή η ρήτρα. Επίσης, να σα ότι όταν διαπραγματευθήκαμε τον Ιούνιο, αυτό το οποίο είχε μπλοκάρει αυτή τη συμφωνία. Ήταν αυτός ο λόγος, γι' αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο έγινε εσφεσμένη αυτή η συμφωνία τον Ιούνιο, γιατί είχε καθυστερήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. μέχρι τούδε υπήρχε μια μεταβατική συμφωνία, η οποία ίσχυε και βεβαίω. Και βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι το θέμα της ελληνίας πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα και στη συμφωνία και η λύση την οποία είχαμε βρει τότε, τον Ιούνιο δηλαδή, ήταν να εξασφαλίσουμε αυτή τη συνεχή ροή, γιατί αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα που είχαμε θέσει όσον αφορά την ελήψη στα ύδατα τη χώρα αυτή. Η διαπραγμάτευση λοιπόν βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν θα ήθελα να περάσω αυτή τη στιγμή σε περισσότερε λεπτομέρειε, αλλά έχουμε κατά νου αυτή τη στιγμή μια συμφωνία η οποία θα είναι πολύ πιο μακροχρόνια, τριετή δηλαδή. Οι διαπραγματεύσει λοιπόν βρίσκονται σε εξέλιξη πριν λίγες εβδομάδες είχε γίνει συνεδρίαση παρήφη των θεμάτων αυτών, υπάρχουν τα πρακτικά και ένας δεύτερος κύκλος θα γίνει το ε, Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, πάλι στις Βρυξέλλες η οποία αυτή η συνάντηση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί. Ε, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, αλλά θα γίνει. Σκοπός μας είναι αυτή τη στιγμή να περατώσουμε αυτή την όλη διαδικασία την 15η Μαρτίου. Είναι κάτι το οποίο ήταν γεγραμμένο στο προηγούμενο πρωτόκολλο. Υπάρχει δηλαδή προθεσμία και πρέπει να πετύχουμε μέχρι τη 15η Μαρτίου και θα πρέπει βεβαίω εν ευθέτω χρόνο να έχει οθετηθεί για να τα πράγματα να εξελιχθούν κανονικά. Τώρα έρχομαι σε θέματα τα οποία άφτονται, είναι πιο συγκεκριμένα μάλλον. Η κυρία Ντεβίνια έθεσε όσον αφορά αυτή τη συμφωνία, στο, αναφερόμενη αυτή στο άρθρο 5 και τη δυνατότητα να επανεθεωρηθεί το θέμα της αλληλείας. Το άρθρο αυτό, ξέρετε, άπτεται πάντοτε του, αυτή, του αυτού κονδυλίου του προϋπολογισμού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Βέβαια στο θέμα αυτό δεν τίθεται πλέον καθότι η υπόθεση αυτή είναι εντελώς θεωρητική και έχουμε μέχρι ένα χρόνο ακόμη για την περάτωση, για, την, για τη λήξη αυτής της συμφωνίας και βεβαίως μέσα σε αυτό το χρόνο θα υπάρχουν δυνατότητες για τις, θα επιλεγούν εκείνες τις δυνατότητες οι οποίες δίνονται μέσα από αυτή τη συμφωνία. Το ίδιο ισχύει και σε αυτό το οποίο τίθεται ε, για το άρθρο 6.5 6.5 για τα ψάρια, τα απορρίμματα των ψαριών είναι τεχνικά θέματα τα οποία τα εξετάζουμε και θα τα επανεξετάσουμε βεβαίως ε, με το θέμα της επαναδιαβάτευσης της όλης συμφωνίας. Επίσης, το θέμα αυτό που είπατε, ποιες είναι οι μη κανονικές συνθήκες, ανώμελες συνθήκες, εκτός ε, μη φυσικές ε, αυτές θεωρούμε εμείς μια ε, ε μαύρη ε, καταστροφή η οποία μπορεί να γίνει από πετρέλαιο και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο που μπορεί να διακοπεί πλήρως η αλίευση ε, όπως είχε γίνει πραγματικά με, τις, με τον Σαλωμόν με το Σολομό, συγγνώμη. Ξέρετε, μια ολόκληρη περιοχή, λόγω αυτή τη διαρροή του πετρελαίου, είχε, μια ολόκληρη περιοχή είχε απαγορευτεί στην ελίευση. Έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι έχουν εγγραφεί μέσα σε αυτή την υποέγκριση συμφωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εφόσον έχει απαντήσει η Κομισιόν σε όλα αυτά, όσον αφορά τη δυνατότητα για το ποσοστό εκείνο το οποίο θα πρέπει να αλλιεύεται στο μέλλον. Οποιαδήποτε απόφαση η οποία θα πρέπει να ληφθεί θα πρέπει να βασίζεται, θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και χαίρομαι πάρα πολύ ότι η Κομισιόν επιμένει σε αυτό το θέμα και το έχει γράψει μέσα σε σχέση με τη συμφωνία. Αλλά γενικότερα θα ήθελα να πω υπήρξαν θετικές απαντήσεις από τους άλλους συναδέλφους σε αυτή την ατζέντα και για το, θέμα, για, το, για το θέμα αυτό και οι επιτροπές του προπολογισμού και άλλες επιτροπές δώσαν θετική, ε, θετικό ok. Έτσι λοιπόν είμαι πάρα πολύ ευτυχής να λάβω υπόψη μου οποιαδήποτε σχόλιο το οποίο θα έρθει και το οποίο πραγματικά μπορεί να εισαχθεί και σε μια οποιαδήποτε τροπολογία σε αυτό το θέμα. Για να δείξει πραγματικά ο καθένας τη δική του διάθεση να τα έγραψε αυτά. υπάρχουν επίση αυτέ οι δυνατότητε που δίδονται όσον αφορά τη δεξιευτή. Σα ευχαριστώ πολύ. Όλοι συμφωνούμε λοιπόν από ό,τι βλέπετε κύριε Χακλούντ και περνάμε τώρα στο χρονοδιάγραμμα σχετικά. Η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης ε, είναι σήμερα, έτσι, 19 Δεκεμβρίου. Για την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 6 Ιανουαρίου, μεσημέρι 12.00 και θα ψηφίσουμε προς έγκριση στην συνεδρία 24 και 25 Ιανουαρίου 2012. Καταρχήν προβλέπεται ότι θα πάει στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου προς έγκριση στην Ολομέλεια. Και έτσι κλείνουμε το σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη του κυρίου Χάγκλον. Σας ευχαριστούμε κύριε Χάγκλον. Περνάμε στο 5. Τροποποίηση του κανονισμού 1967 κάθετος 2006 του Συμβουλίου σε σχέση με τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο. Η συγκήτρια κυρία Ρόσμπαχ. Ήδη κατά την τελευταία συνεδρίαση είχαμε μια παρουσίαση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτής της πρότασης που είναι μια προσαρμογή και εξίσωση των ε, ρυθμίσεων για την επιτροπολογία του νέου κανονισμού σε ισχύ και έπρεπε και πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα επιτροπολογία ως διαδικασία μετά τη συνθήκη Λισαβόνας. Γι' αυτό δίνω τον λόγο στην κυρία Ρόσμπαχ για να μας εκθέσει την άποψή της. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε κι εσείς, πρόκειται για μια νέα διατύπωση την οποία θα πρέπει να έχουμε προκειμένου να καταφέρουμε να τονίσουμε τις νέες αρμοδιότητες που προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για τον πρώτο κανονισμό που έχουμε όσον αφορά τα αλλιεύματα, του λευτικούς πόρους στη Μεσόγειο θάλασσα, για τον πρώτο κανονισμό ο οποίος πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις νέες αρμοδιότητες που προβλέπονται. Ήδη έχουμε ένα έγγραφο διαθέσιμο. Αλλά βέβαια θα προκύψουν και κάποιες ερωτήσεις και ήδη έχουν υποβληθεί κάποιες ερωτήσεις από τη δική μας την Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι το όλο εγχείρημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά βέβαια έχουμε ήδη εντοπίσει κάποιες ε, δυσκολίες στην πρώτη φάση. Για παράδειγμα, πρέπει να καταφέρουμε να πετύχουμε την κατάλληλη ευθυγράμμιση όσον αφορά τους κανονισμούς που άπτονται της αλίας και πρέπει να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση προκειμένου να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα της νέας αρμοδιότητας που προβλέπονται από τη νέα συνθήκη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. η κοινή αλλιευτική πολιτική βρίσκεται ακόμα υπό εξέλιξη, υπό επεξεργασία και επομένως δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να βρούμε μία πρωτότυπη λύση εμείς ή αν θα κάνουμε απλώς μία επικάλυψη εργασίας αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η ε, κοινή αλληλευτική πολιτική, η πρόταση κοινή αλληλευτική πολιτική, προκειμένου να αποφύγουμε αλληλοεπικαλύψει. Γιατί καταλαβαίνω ότι ορισμένα πράγματα μπορεί να τροποποιηθούν στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Προφανώ εμεί μπορούμε να κάνουμε την ευθυγράμμιση που προβλέπεται εδώ. Δεν ξέρω όμω αν θα έπρεπε να περιμένουμε, γιατί αν κινηθούμε κι εμεί παράλληλα, μπορεί να προχωρήσουμε σε αλληλοεπικαλύψει. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι και μόνοι σας μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο και να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Επί της αρχής, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε αν το παράρτημα αυτό από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι γενικόλογο, είναι ιδιαίτερα αόριστο, ή αν θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ε, ε, αλλαγές στην διατύπωση, για παράδειγμα να λέγεται the institutions, τα θεσμικά όργανα, ή αν θα πρέπει να γίνονται σαφείς αναφορές στις πράξεις κατεξοδότηση και στις εκτελεστικές πράξεις, εκεί δηλαδή που προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί μόνη της να παίρνει κάποιες αποφάσεις. Ίσως στις περιπτώσεις αυτές να πρέπει να δούμε αν εμείς θα είμαστε σε θέση να επιτηρούμε τις αποφάσεις αυτές που θα ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βλέπετε ότι στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής δεν ρωτούνται τελικά τόσο πολύ τα κράτη-μέλη. Εν τέλει μπορεί να είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η οποία θα αποφασίζει εξ ονόματος των κρατών μελών όσον αφορά την αλία στη Μεσόγειο θάλασσα. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει κάποια στιγμή αργότερα μία συζήτηση εκ νέου, όταν θα έχουμε και το τελικό έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένω θα, θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο στη συνεδρίαση που προβλέπεται για το Φεβρουάριο. Τέλη Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθο, θα έχουμε το τελικό έγγραφο. Ίσως τότε λοιπόν να πρέπει να γίνει συζήτηση. Δεν ζήτησε κανεί τον λόγο. Θα ήθελα όμω να εκφράσω μια άποψη εγώ προσωπικά. Πιστεύω, κυρία Ρόσπαχ, εγώ ότι σε αυτή την περίπτωση εμείς πρέπει να προσαρμόσουμε τον κανονισμό στη νέα επιτροπολογία μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η παλαιά τροπολογία ως διεργασία είναι ανεδαφική, έχει ξεπεραστεί. Και σε σχέση με τους κύριους κανονισμούς έχουμε την υποχρέωση να προσαρμόσουμε τώρα εμείς τις διεργασίες στη νέα διαδικασία επιτροπολογίας. Δεν υπάρχει άλλη ε, πορεία από το να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Εγώ τις προάλλες έχοντας δει αυτή την πρόταση και έχοντας υπάρξει ως εισηγήτρια, έχοντας λειτουργήσει ως εισηγήτρια για τον κανονισμό στον παρελθόν, συμφωνώ καταρχήν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή για τις προτάσεις που γίνονται κατεντολήν, με κατεντολήν πράξης, ε, ωστόσο με μια εξαίρεση που είναι τα παραρτήματα και κυρίως για το παράρτημα για τις ελάχιστες διαστάσεις. Και σε σχέση με τα παρατήματα, ειδικά για τα παρατήματα, ιδιαίτερα όμως για τις διαστάσεις, το παράτημα για τις διαστάσεις και για τα θέματα τα οποία είχαν δημιουργήσει τριβές ε, όσον αφορά τον, την διαπραγμάτευση του κανονισμού όσον αφορά τεχνικές λεπτομέρειες είναι ένα θέμα που πρέπει να παραμείνει σε συναπόφαση και όχι σε κατεντολήν πράξης. Για τις υπόλοιπες προτάσεις θεωρώ ότι είναι σωστές από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκονται στην ίδια γραμμή πλεύση για την επιτροπολογία όπω και στον προηγούμενο κανονισμό. Απλά τώρα προσαρμόζονται στι νέε ε, αποφάσεις και ρυθμίσει για την επιτροπολογία, εν πάση περιπτώσει. Εγώ όμω σας λέω ότι πρώτον, <clears throat> σε σχέση με την ερώτησή σας, πιστεύω ότι πρέπει να προσαρμόσουμε αυτό στην νέα επιτροπολογία. Δεύτερον, σύμφωνο με την πρόταση της Επιτροπής για τις κατεντολήν πράξεις για τα διάφορα άρθρα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω όλα αυτά, αλλά με εξαίρεση τα παρατήματα. Τα παρατήματα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με τι ελάχιστε διαστάσει, το θέμα αυτό θα ήθελα να το εξαιρέσουμε και για τα παρατήματα που μπορούμε, πρέπει να εξαιρέσουμε. Αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε για τα παρατήματα. Αυτά σε σχέση με την ε, εξέταση ανάρθρω, με την παλαιά τροπολογία όπως ίσχυε που ε, τώρα προσαρμόζεται, πρέπει να προσαρμοστεί. Συμφωνώ λοιπόν να προσαρμοστεί η πρόταση της Επιτροπής ως έχει με εξαίρεση αυτή τις λεπτομέρειες που σας εξήγησα και που πρέπει να συζητήσουμε σε περισσότερο βάθος. Συμφωνώ λοιπόν να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε με την πρόταση ως έχει, με εξαίρεση, όπως είπα και εμένω και επιμένω, με εξαίρεση τα παρατήματα. Λοιπόν, από πλευρά τη Επιτροπής παρακαλώ, εσείς κύριε Χρυδόν Λόγκ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ θετική ανταλλαγή απόψεων που είχαμε για το ζήτημα αυτό. Ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική αυτή η ανταλλαγή απόψεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ίδιο ελπίζω και για την εισηγήτρια. Είχαμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε περισσότερο σε κάποια ζητήματα τα οποία είναι τεχνικά και όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε πρόκειται για ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με τις θεσμικές διαδικασίες, δηλαδή αυτές που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να εφαρμοστεί ένα μηχανισμό λήψη αποφάσεων ο οποίο να συνάδει με την κατάσταση όπως έχει στη Μεσόγειο, από την άλλη όμως ενδεχομένως να, διαφορε... να υφίστανται διστάμενες απόψεις όσον αφορά τον κατάλογο τροπολογιών που προβλέπεται όσον αφορά τι ε, κατεξοδότηση πράξη ή τις ε, αποφάσεις εκεί πέρα που μπορούν να ληφθούν με συναπόφαση. Όσον αφορά τώρα την ε, σημασία του να καταφέρουμε να αποφασίσουμε για την πρόταση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της σε συνεργασία με τα περισσότερα κράτη-μέλη της Μεσογείου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι ο κανονισμός αυτός ο οποίος έπρεπε να αρχίσει να ισχύει πλήρως το 2007 και του οποίου η μεταβατική φάση ολοκληρωνόταν το 2010 για ορισμένα άρθρα, προκειμένου λοιπόν ο κανονισμός αυτός να μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως και να τηρηθεί πλήρως από τα κράτη-μέλη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ορισμένες διατάξεις ε, της πρότασης αυτής είναι διατάξεις που από τις αρχές του 2012 θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσω του λευτικού τομέα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα να αποφασίσουν για τους μηχανισμούς εκείνους που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αποκριθούμε στις, στα αιτήματα τα οποία προκύπτουν από τον κανονισμό αυτό. Πραγματοποιήσουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε γρήγορα, ξεκάθαρα ποια είναι η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώ επίση και ποια είναι η στάση του Συμβουλίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσουμε για ένα ξεκάθαρο μηχανισμό λήψη αποφάσεων. Επ' αυτού λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθεί γρήγορα μία απόφαση, πέρα από τι άλλε συζητήσει που θα μπορούσαν να γίνουν για πιο συγκεκριμένα άρθρα. Πάλωστε δεν συζητάμε αυτά σήμερα. Συμφωνώ λοιπόν με αυτά τα οποία είπατε όσον αφορά τη δυνατότητα, μιας, τη δυνατότητα λήψης μιας απόφασης πολύ γρήγορα, γιατί όπως εξήγησα ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο γρήγορα, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε έναν γρήγορο διαφανή μηχανισμό για όλους τους φορείς, από τους ιδιωτικούς φορές που θα το χρησιμοποιήσουν μέχρι τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χρειαζόμαστε επίσης και ένα μηχανισμό λήψης αποφάσεων, πιο συγκεκριμένα για τα ζητήματα λία στην Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ισηγήτρια, θέλετε να προσθέσετε κάτι ή μπορούμε να προχωρήσουμε στο χρονοδιάγραμμα. Θέλετε να πείτε κάτι, όχι, τέλεια. Λοιπόν, θα καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα τώρα. Ως εξής, ε, παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης ε, προβλέπεται για τις, ε, την 28 Φεβρουαρίου ψήφιση προς έγκριση στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή 21 Μαρτίου και θα περάσει στην Ολομέλεια της περίοδου Συνόδου του Απριλίου. Έτσι με αυτά ευχαριστώ τον κύριο εισηγητή Ντονατέλα για την ε, παρέμβαση αυτή. Περνάμε στο 5 για την υπομονή του, περνάμε στο 6 για την ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Η συγγήτρια είναι η κυρία Λέβιν. Δίνω τον λόγο λοιπόν στην εισηγήτρια ευθύ αμέσω ε, την κυρία Λέβιν. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. <clears throat> Thank you, Madam President. Uh, yes, I get... Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι έχετε διαβάσει την ανακοίνωση που έχει δοθεί εκ μέρου τη Κομισιόν για την εξωτερική πολιτική τη ΕΕ. Όπω γνωρίζετε λοιπόν, η ΕΕ είναι μία από τις λίγους από τους λίγους παγκόσμιους πρωταγωνιστές σε όλο τον κόσμο και είναι αυτή η χώρα που έχει διμερείς συμφωνίες, έχει μεγάλο στόλο κλπ. Και νομίζω πως ε, και υπάρχει μια οργάνωση τεράστια γύρω από το θέμα αυτό. Επίσης είναι από τους βασικούς, από τους βασικές αγορές για την παραγωγή και την κατανάλωση εισάγουμε το 25% των αλλιευμάτων του κόσμου. Ένα στα τέσσερα ψάρια είχατε στην Ευρώπη λοιπόν και αυτό μας δίνει με τεράστιες ευθύνε στην Ευρώπη και για την ΕΕ να δεσμευτεί όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς επίσης και τη συντήρησή της των ελευμάτων δηλαδή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η δέσμευση θα πρέπει να πάει λίγο παραπέρα πέρα από τη σημαντική στο ΦΑΟ και άλλους οργανισμούς με τις διμερείς συμφωνίες κλπ. Μερικές από αυτές τις ε, οι ιδέες είχαν ήδη αναπτυχθεί πριν δύο μήνες σε μια έκθεση η οποία κατέθηκε αυτό το θέμα και ποιος θα ήταν ο ρόλος του ΕΕ για την καταπολέμηση αυτής της καταστάσεως που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν ακόμη και πώς πραγματικά αυτή τη στιγμή να λάβει την πρωτοβουλία για τη συντήρηση καθώς και την προώθηση τη της και θα προσπαθήσει επίσης ένα ένα πεδίο στο οποίο θα μπορούν πραγματικοί όλοι οι παίκτες οι οποίοι και συμβαλόμενοι να μπορούν να παίξουν το σωστό παιχνίδι, ιδιαίτερα σε αυτές τις ε, ποσότητες που εισάγονται στην ΕΕ. Γιατί αυτή η ευθύνη της ΕΕ υπάρχει μία μεγάλη ευθύνη για όλους εκείνους τους στόλους οι οποίοι δρούν και αναπτύσσονται εκτός της μέσα μέσω ιδιωτικών επενδύσεων που γίνεται σε αυτό το θέμα. Επίσης θα πρέπει να δούμε πραγματικά τι είναι εκείνη η ε, κερδοφόρα επιχείρηση η οποία βρίσκεται, ποια είναι, τι συμφέροντα κρύβεται πίσω από αυτό. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να βρούμε πώς μπορούν να υπάρχουν διαφυγέ, πώς μπορούν να υπάρχουν λύσεις για αυτό το θέμα και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά υπάρχουν όλο και περισσότερα έτοιμα εκ των πολιτών για το θέμα της βιωσιμότητας αυτής της δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο στις συμφωνίες οι οποίες υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο δράσης για όλους τους ε, συμμετέχοντες σε, αυτή την, σε αυτό το χώρο. Επίσης και ένας στόλος ο οποίος θα πρέπει να συμμετέχει θα πρέπει να έχει μια λογική, δηλαδή θα πρέπει να βάζουμε ποσοστό όσον αφορά τις, ε, τα εισαγόμενα ψάρια τα οποία βέβαια αυτά τα εισαγόμενα ψάρια βγαίνουν εκτός των ποσοστών των συμφωνιών. Επίσης θα πρέπει να δούμε κάτι το οποίο ε, το Γενάρη θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, 23-24 Γενάρη για αυτό το θέμα εδώ και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Αλλά σήμερα θα εστιαστώ μόνο στο πιο σημαντικό, το οποίο είναι μέσα στην ανακοίνωση της, ΕΕ, της Κομισιόν για την εξωτερική πολιτική, για τη συμμετοχή την οποία θα πρέπει να υπάρχει όσον αφορά τον ελευτικό τομέα και, και λέγονται ότι είναι βιώσιμα, καθώς ε, επίσης σε μια πολιτική στα πλαίσια της ΦΑΟ, η οποία θα πρέπει να είναι πολύ πιο μακροχρόνια Ξεκινάω όμω από αυτό το τελευταίο θέμα. Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει διμερής διάλογος με τους εταίρους μας, πράγμα το οποίο είναι σημαντικότερο και πολύ κρίσιμο. Επίσης μια, ε, μια προσέγγιση του οικοσυστήματος συστήματος ολόκληρου με βιώσιμη δυνατότητα και σφαιρική αντιμετώπιση. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό πράγμα και νομίζω πως πραγματικά έχει τεράστια ευθύνη η Κομισιόν σε αυτή τη διαδικασία και τον, τον λόγο τον οποίο θα αναπτύξει. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει, όπως λέγεται, συνεργασία με τους βασικούς εταίρους και αυτό είναι καταπληκτικό. Τα, κύματα, τα κείμενα αυτά τα οποία υπάρχουν και μια γενικότερη αρχιτεκτονική όσον αφορά την αλληλεία είναι κάτι το καταπληκτικό και το οποίο θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια της εθνικής δοσιδικίας για την επίλυση των προβλημάτων τα οποία ε, ανακύπτουν. Και αυτό είναι επίση κάτι καταπληκτικό. Αφετέρου τώρα υπάρχει κάτι με το της ανακοινώσεως της οποίο με αφήνει αρκετά σκεπτική και θα ήθελα να οθήσω την Κομισιόν να είναι πιο σαφή σε αυτό. Θα είναι η πρόταση τη βασικών εκείνων προτάσεων που θα γίνουν όσον αφορά εκείνη την προσπάθεια που γίνεται για την, για την ποσότητα εκείνη των ελευμάτων η οποία θα πρέπει να μειωθεί. Ξέρετε, δεν υπάρχουν σε αναπτυσσόμενες χώρε και σε παραπτικές χώρε τέτοιες δυνατότητε να αγοράσουν τέτοιες ποσοστώσει. Και καταλαβαίνετε υπάρχουν ε, μερικά τα οποία είναι εντελώς ξεπερασμένα και δεν πρέπει να βρίσκουμε σε αυτή την έκθεση. Επίση. οι απόψει που σε αυτών των διαφόρων οργανώσεων είναι πάρα πολύ σημαντικέ, δίνουν πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία ε, ε, Επίσης, τα συμβαλόμενα μέλη είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια περισσότερη δεσμευτική προσπάθεια των συμβαλωμένων μερών για την ανάληψη αποφάσεων, πολύ καλύτερα από αυτή που υπάρχει σήμερα, αλλά η αποφαστική διαδικασία ε, να μην γίνεται μια συμφωνία η οποία δεν συνάδει με τους ήδη υπάρχοντες κανόνες. Ερχόμενο στο, στο μέλλον όσον αφορά τη βιωσιμότητα των συμφωνιών, αυτό που αποκαλείται έτσι και νομίζω Νομίζω πως υπάρχουν πάρα πολύ καλές αρχές οι οποίες έχουν γραφεί μέσα στην ανακοίνωση αυτή. Η αναγνώριση ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, ε επιστημονικοί έλεγχοι οι οποίοι θα γίνονται εκ των προτέρων πριν καθομολογηθεί η συμφωνία καθώς επίσης ε, αυτά τα οποία λέγονται και άλλα πολλά εδώ, νομίζω πως πραγματικά αν δεν μείνουν στα λόγια και δεν είναι ωραία λόγια, είναι πολύ καλά πράγματα αυτά τα οποία προτείνονται. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια δυνατότητα διαφάνειας για το σύνολο των λεωμάτων από τους τοπικούς και τους ξένους και άλλους οι οποίοι συμμετέχουν. Νομίζω πραγματικά ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εξέταση η οποία θα πρέπει να γίνεται εκ μέρους επιστημονικών ομάδων οι οποίοι θα παρακολουθούν ιδιαίτερα στη Δυτική Αφρική όπου θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις και αναλύσεις γι' αυτό. Το θέμα της διαφάνειας σημαίνει ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί και η διαφθορά η οποία υπάρχει και σε αυτό το μέρα των μη κυβερνητικών κυβερνήσεων τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης συμφωνούμε με την πρώτη Κομισιό ε, για το διαχωρισμό των δύο τομέων Εάν αυτή τη στιγμή ότι μειώνονται ο, τα, ε, αποθέματα των κυπόροι οι ελευτικοί, δεν αδικαιολογείται αυτό το πράγμα ότι, ότι, ότι αυτό θα, θα πρέπει να μείνει άμυρο στην προσπάθεια εκείνη που γίνεται με όλες εκείνες τις συμφωνίες οι οποίες από το τομέα αυτού και εκείνο και με άλλες χώρες ότι δεν θα πρέπει βεβαίω να χρηματοδοτείται εκ μέρου των φορολογημένων μια τέτοια πολιτική. Όσον αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι εκ των όνων ουκάνευ μια συμφωνία, εφόσον θα πρέπει να εγγράφεται και αυτή μέσα. Και πιστεύω πω η αρχή τη ε, ε, αποκλειστικότητα θα πρέπει να τηρηθεί και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ε, να μην υπάρξει μια φυγή εκ μέρους, των, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Στόλου η οποία έχει ε, σημαία της κοινότητος. Νομίζω πως πραγματικά θα πρέπει να γίνεται πιο μια τακτική ε, επιθεώρηση όλων αυτών των πραγμάτων ε, και εκ μέρους επί της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης. Εάν δεν επιτύχει αυτό, αν έχει επιτευχθεί αυτό επιδιωκόμενο, τότε θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα μια αναθεώρηση των συμφωνιών αυτών για τη βιωσιμότητα πάνω με το πάντοτε των πραγμάτων. Επίσης θα πρέπει να, να δούμε ποιες είναι εκείνες οι προσδοκίε και οι στόχοι και οι φιλοδοξίες των απτυσσομένων εκείνων χωρών γι' αυτό. Έτσι λοιπόν η βιωσιμή αλλιεύση, η θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στην χώρες και στις κυβερνήσεις των χωρών αυτών να έχουν δυνατότητα ανάπτυξης αλλά και να υπάρχει μια βιώσιμη ε, αλληλεία και σε αυτές τις χώρες. Νομίζω πως πραγματική σε αυτές τις δύο πτυχές θα πρέπει να αναλάβουμε τις μεγάλες ευθύνες τις οποίες έχουμε. Όσον αφορά την προθεσμία και την παρουσίαση του σχεδίου, θα γίνει στις τέλος Φεβρουαρίου και οι προθεσμίες 15 Μαρτίου προθεσμία για τις τροπολογίες και βεβαίως θα περάσει τον Απρίλιο. Χαιρετίζω βέβαια εκ των προτέρων και καλωσορίζω οποιαδήποτε, οποιαδήποτε σχόλιο, παρατήρηση κλπ. που θέλει να γίνει από του συναδέλφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε σχέση με την, τα κυριότερα σημεία της ανακοίνωσης τα ανέφερε η κυρία Λεβίν. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι ή πρέπει να είναι η εξωτερική διάσταση στην πολιτική αλληλείας γιατί πρέπει να καθορίσουμε σαφώς τι επιθυμούμε να είναι αυτή η εξωτερική πολιτική. Και αυτό αποτελεί έναν από τους κυριότερους πυλώνες ε, της κοινή αλλιευτικής πολιτικής ε, και φυσικά ισπανικής. Χωρίς αμφιβολία θεωρούμε ότι είναι ένα ουσιώδες, το στοιχείο. Αλλά πέρα από αυτά τα οποία συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα με τη συμφωνία με το Μαρόκο, έχουμε και την ίδια διαπραγμάτευση τώρα τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τη Μαυριτανία. Και είναι η χρονική στιγμή που έχει σημασία κλειδιού για να προβληματιστούμε και να δούμε τι σημαίνει η εξωτερική διάσταση για την κοινή πολιτική αλληλεία και κυρίως ποια συμπεράσματα θα συναγάγουμε σε σχέση με αυτή την πολιτική αλλιευτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Αληθεύει ότι μπορεί να είναι προ όφελο ε, τη ε, κοινότητα ε, να μην μειωθεί αυτή η διάσταση. Αλλά δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην συρρήκνωση του οικονομικού ρόλου. Δεν μπορεί μόνο αυτό να είναι ο ρόλο των διαπραγματεύσεων για τον οικονομικό ρόλο. Και υπάρχει μετά και ένα άλλο θέμα, το οποίο πιστεύω ότι είναι θεμελιώδους σημασία και αυτό. Να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε με την, ας το ενδυνάμωση των ιδιωτικών συμφωνιών που δεν υποβάλλονται στα ίδια κριτήρια ή δεν έχουν τις ίδιες αρχές ε, όπως οι συμφωνίες αλληλείας ε, σε σχέση με τις κοινοτικές συμφωνίες έχουμε μεγάλο κίνδυνο εδώ μπροστά μας που ε, διαγράφεται και πέρα από την ανασφάλεια και αβεβαιότητα που μπορεί να δημιουργηθεί και μετά έχουμε και την υπογραφή νέων συμφωνιών και την αναζήτηση νέων ευκαιριών για την αλληλεία που πρέπει να συνεχίσει να είναι ένα αντικείμενο της εξωτερικής πολιτικής για την αλληλεία. Μεταξύ άλλων για να αποφύγουμε οικονομικές ζημιές, αλλά επίσης να διασφαλίσουμε με αυτόν τον τρόπο μια υφόρο εκμετάλλευση των αλλιευμάτων πράγμα για το οποίο γίνεται συχνά λόγος στην ανακοίνωση. Και κυρίως και η ανάπτυξη της τοπικής αλίας και του τοπικού δυναμικού. Πρέπει να δούμε τις τεχνικές προϋποθέσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα να αλλιεύει ο αλλιευτικός στόλος της κοινότητας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη συμφωνία με την Μαυριτανία. Και φυσικά δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία του να δυσχεραίνονται οι δραστηριότητες των σκαφών και του στόλου σε σχέση με αυτό το θέμα γίνεται λόγος ε, για κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες και δεν αναφέρεται από την ανακοίνωση. Δεν υπάρχουν οι ίδιες απαιτήσεις ε, ελέγχων και εποπτείας όσον αφορά τους αλλιευτικούς πόρους ε, ε, όσον αφορά τα, ε, τις προδιαγραφές που ισχύουν για τον κοινοτικό στόλο. Και σε σχέση με τις ε, προδιαγραφές αυτές είναι απόλυτα αναγκαίο να δούμε ότι δίνουμε μεγάλη, συμφωνία, μεγάλη σημασία σε αυτές τις πτυχές, κυρίως περιβαλλοντικά και θα πρέπει η πολιτική διασφάλισης και συντήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πολύ πιο προστατευτική σε σχέση με την πολιτική που μπορεί να ακολουθηθεί με διμερείς συμφωνίες όσον αφορά τρίτες χώρες χωρίς τέτοιου είδους φιλοπεριβαλλοντικές διατάξεις εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίζουμε τις φιλοπεριβαλλοντικές πτυχές να συνεχίσουμε τον αγώνα κατά της παράνομης αλίας ε, όσον αφορά την ε, πολιτική μας ε, είναι ένα άλλο, μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξετάζουμε πάντα υπό το πρίσμα αυτού που εμείς υπερασπιζόμαστε πάντα, δηλαδή την αηφόρο εκμετάλλευση των αλλιευμάτων. Ένα θέμα που επανειλημμένα αναφέρεται σε αυτή την ανακοίνωση, αλλά που πρέπει πραγματικά να είναι αποτελεσματικό και από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκείνου του είδου ε, τα αλλιεύματα από πλευρά των τρίτων χωρών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το περιβάλλον. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι ε, τοπικέ οργανώσει αλληλεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενδυναμώσει τη δράση τη κατά τη πειρατεία και κατά τη παράνομη αλληλεία. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και πρέπει να συνεργαστούμε όλοι και ευχαριστώ την συγγήτρια για το έργο τη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η γαλλική τηλεόραση, ο σταθμός France 3, ε, το τρίτο κανάλι θα ε, μαγνητοσκοπήσει για μια διάρκεια 10 λεπτών. Να το ξέρετε λοιπόν ότι βρίσκεται εδώ αυτό το τηλεοπτικό συνεργείο. Έχετε εσείς τον λόγο παρακαλώ. Oui, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την ε, Ιζαμπέλα για την εργασία που έκανε, για αυτή την ε, έκθεση πρωτοβουλίας και να φερθώ σε κάποια ενδιαφέροντα σημεία. Πρώτον, η πιο διαφανής και πιο ελεγχόμενη χρήση της ε, κοινοτική χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, περαιτέρω ανάπτυξη επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και αυτό πολύ σημαντικό. Μηχανισμοί εποπτείας όσον αφορά την ε, κερδοφορία των ε, κρατών που συμμετέχουν στις ε, συμφωνίες αλίας και κάτι ακόμα να μην γίνεται καταχρηστική χρήση των σημαίων όσον αφορά τα αλλιευτικά σκάφη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσα βέβαια να προτείνω και κάποιες τροπολογίες, αλλά θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις πρώτα στην Ιζαμπέλα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να γνωρίζω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνδέσει την εμπορική πολιτική, την ε, σφαιρική εμπορική πολιτική με την ε, πολιτική ελίας, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική αντίφαση ανάμεσα στην, ε, στις παρεκκλήσεις που προβλέπονται, όπως για παράδειγμα για τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα για την Γουινέα Μπισέα, στην οποία αναφερθήκαμε πριν από λίγο, και άλλου κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν για την κοινότητα. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η στάση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μην αλλιεύονται μόνο τα πλεονάσματα αλίας όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες αλίας, αλλά πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα και θα πρέπει να υπάρχει και η χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας. Το ερώτημα λοιπόν που θέτω είναι το ακόλουθο. Προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει γρήγορα με και έρευνα προκειμένου να μην τέθουν εν κινδύνο οι υφιστάμενες συμφωνίες. Και κάτι ακόμα, το οποίο ακούσαμε και πριν από λίγο, θα θυμάστε πώς εξελίχθηκε η ψηφοφορία την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά τη συμφωνία με το Μαρόκο, την επέκταση που προβλέπετε εκεί. Πολλοί είναι υπέρ της αλληλευτικής αυτής συμφωνίας με το Μαρόκο, αλλά την απέρριψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συμφωνία αυτή εφαρμόστηκε με προσωρινό τρόπο, αναμένοντας την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι αλλιευτικοί φορείς στα σκάφη τα οποία λείπαν στα νυχτά του Μαρόκου. Όπως το γνωρίζετε χρειάστηκε να αποσυρθούν από τα ύδατα αυτά του Μαρόκου. Ουσιαστικά τους διώξαμε από την περιοχή. Το ερώτημα που θέτω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το ακόλουθο. Αυτό ουσιαστικά θέτει αν κινδύνω την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας όπως προβλεπόταν για το Μαρόκο και γενικότερα μέσω της ψηφοφορία αυτής δημιουργείται προηγούμενο θα έχουμε μια νέα νομολογία. Ουσιαστικά αυτή είναι η ανησυχία την οποία εκφράζω. <coughs> Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λόβε για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Έχω πάρα πολλέ ερωτήσει να κάνω, ωστόσο θα κάνω μερικές. Στι προηγούμενες δόσει θα μπορεί να υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο θα δοθεί και τις ιδέες αυτές τις οποίες υπάρχουν για αυτό το θέμα. Δύο σχόλια θα κάνω. Το πρώτο άπτεται στο ρόλο στο εθνικό επίπεδο της Ευρώπης. Νομίζω πως πραγματικά, εάν θέλουμε να κάνουμε πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να, δράσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε όλο τον κόσμο, νομίζω θα πρέπει να ακολουθήσει πολλά αποτελέσματα τα οποία έχουν ε. διότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πολιτική εξωτερική της αλίας. Εάν αυτό θα μπορούν και θα μπορούν να υπάρχουν, αφού είναι πολλές σχέσεις. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένα ολόκληρο κείμενο το οποίο θα πρέπει να υπάρξει για την αλληλεία, πολύ συγκεκριμένα πώς μπορεί να υπάρξει ένα τρόπος και μια έδρα ε, σύμφωνα με την οποία και μερικές αρχές θα πρέπει να γίνεται η πολιτική αιλία σε όλο τον κόσμο. Ένα άλλο θέμα στρατηγικό για τον διεθνή ρόλο της ΕΕ και της πολιτικής της Ευρω... στην Ευρώπη είναι η παράνομη αλλία. Πιστεύω πραγματικά ήρθε η ώρα για να υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα είναι δεσμευτική. Παγκόσμια. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να είμαστε όμως τόσο παθητικοί στις πολιτικές εκείνες οι οποίες γίνεται όσον αφορά τη σύλληψη των παρανόμων εκείνων και της παράνομης αλίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πως αυτές οι χώρες οι οποίες παραβιάζουν θα πρέπει να είναι στο δικό μας χώρο και να συμφωνήσουμε Μπορούμε να αφήσουμε όλες τις υπόλοιπες χώρες απ' έξω, αλλά για την Ορβηγία, για παραδείγματος, 90% εκπροσωπεί του, ε, του ποσοστού εκείνη το οποίο θα πρέπει να, σε, να αυτή την περιοχή. Επίσης, θα πρέπει πάντοτε να εισάγουμε σε οτιδήποτε στη βιωσιμότητα. Δεν σημαίνει βεβαίω τίποτα, διότι έγινε μια πιπίλα αυτή τη στιγμή και είναι μια λέξη που τη βάζουμε ε, ε, τη βάζουμε πάλι, μια είναι της Wikipedia θα λέγαμε, αλλά κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει, διότι το θέμα της βιωσιμότητας δεν είναι μόνο περιβαλλοντολογικό θέμα, είναι το θέμα αυτό, βιωσιμότητα, άπτεται και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Αλία. Και όσο με αφορά, δεν ξέρω πραγματικά αν αυτό το τελευταίο θέμα είναι πρώτο ή δεύτερο, ποιο είναι το πιο σημαντικό, η βιωσιμότητα των εργαζομένων ή του περιβάλλοντος. Δεν το ξέρω ποιο είναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι των εργαζομένων. Είναι λοιπόν το θέμα αυτό της βιωσιμότητας ή ε, θέμα που άπτεται των δικαιωμάτων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω πως στην Κομισιόν έχουμε κάνει διάφορες προτάσεις, αλλά υπάρχουν διάφορες μέθοδοι εντός των οποίων μπορούμε να οικοδομήσουμε τους όρους εκείνους για τη δυνατότητα που μας δίνεται αυτή τη στιγμή για να διακοπεί μια έκθεση η οποία δεν έχει το, πορεία αυτή που θα θέλαμε. Γιατί θα πρέπει να λέμε ότι υπάρχει μια συμφωνία και υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία. Μπορεί να υπάρχει, να υπάρχει, μπορεί να, να, ε, να ανασταλεί, μπορεί να μειωθεί, μπορεί να διακοπεί. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πολιτική αλληλεία προ το ευρώ, δεν υπάρχει το άσπρο μαύρο μόνο. Οι σχέσει οι οποίε υπάρχουν και οι σχέσει όσον αφορά στο, στο τομέα μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε εμά να καθορίσουν όλε τι σχέσει οι οποίε έχουμε με την κυβέρνηση τη απέναντι πλευρά και εμεί να έχουμε τι ευθύνε εκείνε οι οποίε θα πρέπει να αναλάβει και προ αυτή τη χώρα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο, θα πρέπει να σταματήσει αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζεται σε αυτό το τομέα και ξέρετε υπάρχει χώρο που δεν συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία αλλά είτε περάσει είτε δεν περάσει νομίζω ξέρετε ότι θα μπει θα μπει σε υπόμνηση κάπου σε ένα ντουλάπι και κανείς πραγματικά δεν θα ασχολείται με αυτό το πράγμα. Εφόσον βεβαίω μόνο στην περίπτωση που θα γίνει η εκ μέρου Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν, θα πρέπει όχι μόνο να υπογράφει τη συμφωνία, αλλά θα πρέπει να το, να το χειρίζεται κανείς, να το παρακολουθεί, να υπάρχει μια διαχείριση αυτής της συμφωνίας που γίνεται. Έτσι λοιπόν θα πρέπει μέσα στα τριετή αυτή η πορεία ότι θα παρακολουθείτε και εν τη εξελίξη της αυτής συμφωνία η οποία έχει γίνει θα μπορεί να διορθώνεται, να αλλάζει, να επισκευάζεται να το πω έτσι για να δούμε πραγματικά ποια είναι εκείνα τα δικαιώματα τα οποία υπάρχουν. Μπορούμε να τις αγάγουμε αλλά δεν αυτή τη στιγμή, αν το εισαγάγουμε και δεν υπάρχει μια εκτίμηση, μια αποτίμηση τη όλη προσπάθεια που γίνεται, μπαίνει όπω σα είπα προηγουμένω. Και μόνο όταν συμβεί κάτι, αν συμβεί κάτι έκτακτο βεβαίω και πάρα πολύ κρίσιμο, παπ, κόπτεται, διακόπτεται αυτή η συμφωνία. Για πράγμα το οποίο έγινε και το, το Μαρόκο αυτή τη στιγμή. Και εγώ σε αυτό το θέμα, ξέρετε πάρα πολύ καλό, ήμουν υπέρ τη αποφάσεω ότι θα πρέπει να διακοπεί. Και δεν ήταν για ε, θέμα νομικό που σε αυτή την πλευρά και άλλους λόγους ο θα αναπτύξω αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, αν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε και να υπάρξει μία συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτόν, θα πρέπει έτσι να δώσουμε προσοχή. Αυτή η λέξη υλοποίησης θα πρέπει να δοθεί ένα νόημα δηλαδή να δώσουμε ένα περιεχόμενο σε αυτή την πολιτική. Και εγώ εννοώ ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Εκείνες οι πολιτικές οι οποίες γίνονται προς το εξωτερικό, εδώ και λίγα, ε, και λίγα χρόνια θα πρέπει να έχουν μία φυσιογνωμία και η οποία βεβαίως θα ε, γράφεται στην εξωτερική πολιτική. Αλλά η εξωτερική αυτή πολιτική φαίνεται ότι δεν επικρατεί. Και έτσι λοιπόν γίνεται μία συζήτηση η οποία άπτεται μια διπλωματία, θα λέγαμε και μάλλον φρονώ λοιπόν αυτή τη στιγμή να βρούμε στοιχεία τέτοια τα οποία οι επιλογέ οικονομικέ οι οποίε γίνονται στι συμφωνίε τέτοιου είδους τσελίες δηλαδή να είναι να ε, ακολουθούν και να συνάδουν πλήρως με τη γενικότερη εξωτερική πολιτική την οποία να υπάρχει μια, ένα είδος όσμωσης μεταξύ των μεν και των Κατά αυτόν τον τρόπο πραγματικά γύρω προς το εξωτερικό θα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιστευτοί. Σταματάω εδώ. γιατί ξέρετε έχουμε και σήμερα και αύριο και βέβαια έρχονται οι γιορτές και θα πρέπει ε, επιφυλάσσομαι όμως τις επόμενες εβδομάδες να ετοιμάσω ένα κείμενο στο οποίο μπορούμε να εγγράψουμε με στην εκθεσή σας και βεβαίως όποιος θέλει μπορεί να το, το το τροποποιήσει. Έχω και πολλές άλλες ερωτήσεις οι οποίες θέλω να κάνω προς την Κομισιό για την έλλειψη της έκθεσης και της ε, της έκθεσης για την παράνομη αλληλεία, ότι αυτά τα σημεία δεν έχουν ε, εγγραφεί. Και με ένα τελευταίο πράγμα το οποίο είναι πολύ γενικότερο. Εμείς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τομείς όπου η Κομισιό Ξέρετε, η Κομισιόν μας δίνει διάφορα κείμενα, μας δίνει ένα κείμενο εξωτερική πολιτική, για επί της ουσίας, διάφορα άλλα. Και βλέπετε όλα αυτά είναι τμηματικά. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, και αυτό είπα και στην Πρόεδρο, ότι θα πρέπει να συντονιστούν και να υπάρχει, να μην υπάρχει αυτή η κατάτμιση. Διότι όταν υπάρχει αυτή η κατάτμιση βρισκόμαστε ενώπιον μια σχιζοφρένεια η οποία επικρατεί. Ξέρετε, κάνουμε ένα πράγμα στην εξωτερική πολιτική, κάνουμε άλλο πράγμα εδώ και βεβαίω ε, τα παίρνουμε εδώ και τα αποφασίζουμε εκεί, αλλά δεν τα εισάγουμε εκεί και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν ανάγκη σε όλους τους κατηδίαν τομείς να αναπτύξουμε αυτή τη φιλοσοφία που θέλουμε, εάν θέλετε να το πω έτσι, αλλά από την άλλη μεριά να υπάρχει ένα συντονισμός, να υπάρχει μία συνοχή, να υπάρχει μία βάση, πράγμα σε οποίο συνάδελφοι προηγουμένω, προηγουμένως, γιατί διαφορετικά αυτή η βάση σημαίνει που λέγω ότι θα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα διαβιβάζεται σε όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Βεβαίως πιστεύω ότι αυτά είναι δύσκολα να σε αυτό το κοινοβούλιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα καταρχήν να ευχαριστήσω την Ιζαμπέλα. Ήταν σαφέστατο νομίζω ότι πολύ προβληματίστηκε και πολλά πράγματα εξέτασε και σκέφτηκε για να συντάξει αυτό το έγγραφό της. Το πιο αποφασιστικό είναι να δούμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Το μέτρο το οποίο εμείς θέτουμε ως γνώμονα και ως πύχη στις δική μας, στις δικές μας προσπάθειες αλίας, είτε φιλοπεριβαλλοντικά είτε στον οικονομικό τομέα συνολικά, πρέπει να είναι πρότυπο. Πρότυπο για την πολιτική που ακολουθούμε με άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλληλεία. Νομίζω δεν μπορεί να μετράμε με δύο μέτρα και σταθμά. Αυτό είναι που είναι σωστό και δίκαιο για μας στην Ευρώπη πρέπει να ισχύει και στις άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Αν πάρουμε αυτό ως κανόνα, στο τέλος θα έχουμε μια λογική συμφωνία που θα συνάψουμε. Εκείνο που είναι πολύ δύσκολο είναι όταν υπάρχει ρύθμιση όλων αυτών εκ Το ότι συζητάμε για το Μαρόκο και τη Μαυριτανία συνδέεται με το ότι πολλά πράγματα δεν ήταν πολύ συγκεκριμένα και δεν ήταν εξειδικευμένα στις ρυθμίσεις τους. Κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το αντέξουμε στο μέλλον. Οικολογικά, οικονομικά και δημοσιονομικά πρέπει οι συμφωνίες να διαμορφώνονται σε τέτοια πλαίσια ώστε να μπορούμε να αντανακλούμε σε αυτές τις δικές μας πολιτικές. Όταν υπήρξαν μαζικές επικρίσεις ε, ότι τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου διαδραμάτιζαν ένα ρόλο. Ναι, σε σχέση με το Μαρόκο εντάξει, να τα συζητήσουμε αυτά, αλλά να τα συζητήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται νομική ασφάλεια. Αυτό τίθεται ως θέμα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε να υπάρχει νομική ασφάλεια και βεβαιότητα ή θα είναι διακηρύξεις και δηλώσεις προθέσεων. Και στο τέλος αν δεν ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα εξειδικευμένα θα καταλήγουμε σε μια χωρίς όρια συζήτηση. Εγώ θέλω να τα καθορίσουμε σαφώς για να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα μια και δεν ζητεί άλλο τον λόγο θα παρεύω και εγώ. Α, η κυρία Γκαρσία Γέρο. Μα συγγνώμη, δεν το είχαμε δει. Συγγνώμη. Η κυρία καρθία Γέρο παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη πρόεδρε γιατί ήταν τελευταία στιγμή απόφαση να παρέμβω που προκλήθηκε ίσως ακριβώς από την παρέμβαση της ε, συναδέρφου που έλαβε τον λόγο πιο πριν. Είμαι υποχρεωμένη ουσιαστικά να πω και εγώ το ίδιο το οποίο είχε εκφραστεί και σε μια προηγούμενη συνεδρίαση. Η συμφωνία αλίας με το Μαρόκο <coughs> δεν είναι με κανένα τρόπο ένα θέμα που να αποφασίστηκε σε σχέση αυστηρά με τα θέματα μόνο της ε, αλληλείας. Είναι μια απόφαση που ελήφθη που σε κάποιους τομείς μπορεί να τίνει ή να θεωρηθεί ότι υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Είναι όμως μια οικονομική, κοινωνική και φιλοπεριβαλλοντική συμφωνία και πρέπει να γίνεται έτσι για εκείνους που αλλιεύουν σε αυτά τα ύδατα και για τους ε, υπηκόους της Δυτικής Σαχάρα και για τους υπηκόους του Μαρόκου και άλλους. Και το να δούμε όλες αυτές τις πτυχές για τους ε, ε, κατοίκους της Σαχάρας από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών όπως επαναλαμβάνεται συχνά σε αυτό τον τομέα και σε άλλους και προσυπογράφω την ε, παρέμβαση προλαλήσαντος συναδέλφου μέχρι πού μπορούμε να προχωρήσουμε όταν ψηφίζουμε ένα θέμα ή εγκρίνουμε ένα θέμα δεν ρυθμίζεται αποκλειστικά με τον τρόπο αυτό και εξειδικευμένο αν λοιπόν σε σχέση με το μέλλον θέλουμε να είναι σεβαστές όλες οι προϋποθέσεις εργασίας για την αηφορία, για το περιβάλλον, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να κάνουμε ένα παιδαγωγικό, μια παιδαγωγική προσπάθεια, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τη συμφωνία με το Μαρόκο υπό αυτό το πρίσμα. Υπό την ίδια έννοια όπως τα κοινωνικά δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα και η διεθνή νομιμότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σε σχέση με την ανακοίνωση της Επιτροπής θα ήθελα να πω δύο λόγια. Θα ήθελα να πω τα εξής. Για το θέμα της παράνομης αλληλείας, εγώ θα ήθελα ειδικά να τονίσουμε το θέμα της, ε, του ρόλου των περιφερειακών οργανώσεων αλληλείας. Και έχω κάποιες αμφιβολίες για τη σημερινή νομοθεσία σε σχέση με τη μη πλήρη συνεργασία κατά της ε, ε, παράνομης αλίας. Πρέπει να είναι απόλυτα σαφές αυτό, ότι είμαστε κάθετοι όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, το οποίο πρέπει να το δούμε επίσης εδώ και έχει και αυτό μεγάλη σπουδαιότητα, είναι το θέμα της πειρατείας. Η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή πρέπει κάπως να αναφερθεί στο θέμα της πειρατείας. Δεν περιορίζεται μόνο στον Ινδικό ωκεανό, ξεπερνά τον Ινδικό ωκεανό και είναι ένα πολύ επίκαιρο σημερινό πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε και στις Σεϊχέλε. Όχι μόνο στον ειδικό όμως, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Γιατί η γενική διαχείριση είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ε, εντάξουμε στις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με μεγαλύτερη συμμετοχή του τομέα αλληλείας. Γιατί αυτός ο τομέας θα πληρώσει και δεν ξέρουμε σε ποιο ύψος μια σημαντική αύξηση όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες. Και αυτό είναι η ερώτηση που θα ήθελα να διατυπώσω για τις περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας και τη συμμετοχή τους. Θα πρέπει να υπάρχει πιο ενεργό συμμετοχή από ό,τι μέχρι σήμερα αυτού του τομέα. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και περνώ στη συνέχεια στο θέμα, στο θέμα όσον αφορά τις ε, δράσεις Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτό ότι θα προαγάγει, θα προωθήσει ένα σύστημα πρόσβασης ε, πληρωμών για τις περιφερειακές οργανώσεις αλίας. Η ερώτησή μου είναι η εξή: διότι όλα αυτά τα λέτε γενικόλογα εσείς. Αυτή η πρόσβαση σε πληρωμέ ε, ή σε συνεισφορέ που προβλέπεται ως μία από τις δράσεις για τις ε, οργανώσει αλίας αποκλειστικά θα στρέφεται στο κοινοτικό στόλο, στους κοινοτικούς στόλους που α, αλλιεύουν σε αυτές τις περιοχές. Είναι μια πρόθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά των περιφερειών, περιφερειακών οργανώσεων αλλίας για όλα τα σκάφη που αλλιεύουν εκεί. Θα ήθελα να μου το αποσαφηνίσετε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήμουν υπέρ του σε σχέση με τις περιφερειακές οργανώσεις αλλίας να υπάρχει η δυνατότητα με ονόματα των σκαφών που αλλιεύουν και όχι μόνο με ποσοστώσεις ε, για συγκεκριμένους στόλους να αλλιεύουν. Για τις συμφωνίες της διμερής, το impact assessment, ε, η μελέτη επιπτώσεων, είναι αρκετά ε, επεξηγηματική, αρκετά σημαντική. Όταν λέγεται εδώ ότι οι πλειοκτήτες θα πληρώνουν περισσότερα ή ουσιαστικά το σύνολο του ποσού για αυτές τις αλλιευτικές συμφωνίες. Θέλω να μου πείτε πώς θα εφαρμοστεί αυτό, διότι σε σχέση με το impact assessment, σαφές σε σχέση με τις συμφωνίες για, για τον τόνο, υπάρχουν συμφωνίες για τον τόνο που πληρώνουν 100%. Δηλαδή 100 ευρώ ανά τόνο που αλλιεύεται για την αντιστάθμιση όσον, αντιστάθμιση όσον αφορά τους πλειοκτήτες π.χ. για τις Σεϊχέλες υπάρχουν, Σεϊχέλες, υπάρχουν και άλλες συμφωνίες αλίας με μικρότερη εμβέλεια. Θα πρέπει να αναλύσουμε αναπερίπτωση το κάθε ε, υπόδειγμα για να δούμε ποιο είναι το κόστος τέτοιων εμπορικών συμφωνιών. Το να προσπαθήσει κανείς το 100% να πληρώνεται, δηλαδή 100 ευρώ ανατόνο, αυτό φαίνεται ότι είναι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τέλος πάντων αυτό θα είναι το τελικό για τους πλειοκτήτες. Θα πληρώνουν αυτά τα ποσά. Πράγμα το οποίο θα είναι εις βάρος ε, της συνεργασίας για την ανάπτυξη με τρίτες χώρες. Αυτά. Αυτά για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μου αποσαφηνίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναπερίπτωση θα εξετάζεται η αύξηση του κόστους ε, ανασυμφωνία ή όχι. Και τέλος, πώς δικαιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια συμφωνία με τη Μαυριτανία να πληρώνονται 20 εκατομμύρια ευρώ για την βοήθεια για την ανάπτυξη και για παράδειγμα στην Κινέα Μπισάου που έχουμε αύξηση σε 2 εκατομμύρια πώς θα δικαιολογήσετε αυτές τις διαφορές που είναι μεγάλες που προέρχονται και απορρέουν από κακές διαπραγματεύσεις ή μη σαφείς διαπραγματεύσεις. Πώς μπορείτε να το δικαιολογήσετε αυτό. Τέτοια ποσά για την ανάπτυξη, για τη συνεργασία και την ανάπτυξη με τέτοιες διαφορές όσον αφορά για παράδειγμα τις συμφωνίες για τον, την αλία του τόνου και όσον αφορά και τις ε, Σεϊχέλες. Πώς δικαιολογούνται όλα αυτά. Θέλω να είναι σαφή αυτά τα θέματα εκ προημίου για να δούμε πώς θα τοποθετηθούμε υστερότερα ως Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριε Ντοκιπέρ, ε, εσείς, ο κύριος εσείς θα αποφασίσετε κύριε Διευθυντά ποιος θα παρέμβει από εσά για αυτά τα θέματα. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Uh, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και έχουμε καταγράψει όλες τις παρατηρήσεις. Το έγγραφο αναφέρεται ξεκάθαρα στις προτεραιότητες πολιτικής. Βέβαια υπάρχουν ακόμα κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν, να ολοκληρωθούν. Κατάλαβα όμως από τις παρατηρήσεις σας ότι ε, εν γέννη πάνω κάτω συμφωνείται και επιβεβαιώνετε ουσιαστικά τις προτάσεις μας. Επομένως, αποτελεί ιδιαίτερη ενθάρρυνση για μας η στάση σας. Αναφερθήκατε σε κάποια ζητήματα, πολλά μάλλον ζητήματα, δεν μπορούμε όλα να τα εξετάσουμε διεξοδικά. Ή έγινε μια αναφορά για τις επιστημονικές αναλύσεις, καθώς επίσης και το πώς μπορούμε να καθορίσουμε τα πλεονάσματα και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε προς αυτό. Κοιτάξτε, γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον ελευτικό τομέα μέσω διμερών διαπραγματεύσεων και στις πολυμερείς συμφωνίες επίσης έχουμε προσπαθήσει να βοηθήσουμε τους εταίρους μας ε, στο ζήτημα αυτό και γι' αυτό το λόγο έχουμε υποστηρίξει τις διάφορες επιστημονικές επιτροπές οι οποίες εμπλέκονται συμφωνίες αυτές. Επίσης, πολλοί ομιλητέ αναφέρθηκαν στο IUU, στην παράνομη λαθρέα αλία και μας είπαν ε, ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε πιο συγκεκριμένες ιδέες αντιμετώπισης. Μα συστηματικά ασχολούμεθα με το ζήτημα αυτό και προσπαθούμε επίσης να προβούμε και σε ad hoc δράσεις κατά της παράνομης αλίας, πέρα από τις γενικότερες πολιτικές οι οποίες προωθούμε. Και σε διμερές επίπεδο ασχολούμεθα με το ζήτημα αυτό με τους στρατηγικούς μας εταίρους και στην πράξη εφαρμόσαμε κάποιες, ε, κάποιες ε, δράσεις. Η ίδια η Επίτροπος, η κυρία Γαμανάκη, ε, σε ερχόμενη σε επαφή με κράτη με τα οποία συνεργαζόμαστε, εφάρμοσε τέτοιες συμφωνίες. Με τις ΗΠΑ, για παράδειγμα, υπάρχει μια συγκεκριμένη συμφωνία για την καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καλύπτονται όλο και περισσότερο οι δράσεις αυτές στα πλαίσια των συμφωνιών που υπογράφουμε. Επίσης, Είπατε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με κάποιες ε, άλλες ρήτρε, οι οποίες θα οδηγούν σε βιώσιμη ε, αλία, στην καταπολέμηση της παράνομης ε, εργασίας. Όλο και περισσότερο ρήτρε αυτές εντάσσονται στις συμφωνίες που υπογράφουμε με τους εταίρους μας. Και όλο και περισσότερο προσπαθούμε να προσελκύσουμε την προσοχή τους στα ζητήματα αυτά. Βέβαια θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το ζήτημα αυτό περισσότερο, προκειμένου να συνάψουμε τις συμφωνίες αυτές. Έχετε δίκιο ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε εμείς οι ίδιοι καταρχάς στη δική μας την αλία πολύ καλούς κανόνες και στη συνέχεια μόνο να εξάγουμε τους κανόνες αυτούς προς τους εταίρους μας στα πλαίσια των συμφωνιών μας. Προφανώς κάτι τέτοιο προσπαθούμε να κάνουμε και συζητάμε όλο και περισσότερο με τους εταίρους μας στα πλαίσια της σύναψης συμφωνιών, ότι θα πρέπει δηλαδή οι βέλτιστοι κανόνες να ισχύουν και στις δύο πλευρές. Και σε αυτό προσβλέπουμε και με τους ε, μελλοντικούς μας εταίρους. Προσπαθώντας να ξεπεράσουμε κάθε φορά τις σχολίε που προκύπτουν από τη μία την άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε πάντα να γνωρίσουμε πόσα αλληλευτικά δικαιώματα έχουν πουληθεί σε άλλους εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές είναι δύσκολο να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες από τους εταίρους μας. Υπάρχουν ορισμένοι ε, εταίροι μας οι οποίοι ενοχλούνται από την εφαρμογή της ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τους λέμε ότι δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτηση, παρόλα αυτά αυτό δημιουργεί πολλές φορές προβλήματα. Στα πλαίσια πάντα των συζητήσεών μας προσπαθούμε σιγά σιγά να εξηγήσουμε όλες αυτές τις ρήτρε ότι είναι πολύ σημαντικές και ότι είναι και για το δικό του συμφέρον. Σαφώς βέβαια υπάρχουν πολλές φορές κάποια συμβαλόμενα μέρη τα οποία μας λένε ναι ότι βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τους ελευτικούς μας πόρους αλλά έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει προκύψει και σε άλλους τομείς πέρα από την αλληλεία όπου βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν ορισμένες χώρες που στοχεύουν περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη και που προσπαθούν ουσιαστικά να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδοτική συμβολή σε κάθε συμφωνία. Προκύπτουν λοιπόν αυτά τα προβλήματα και προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να μειώσουμε την πίεση που ασκείται, την αλληλευτική προσπάθεια η οποία ουσιαστικά βαίνει κατά των αλληλευτικών πόρων, αλληλευτικών αποθεμάτων. Το IUU το έχουμε καλύψει στα πλαίσια των FMOs. Στις συζητήσεις που κάνουμε προσπαθούμε να πείσουμε όλα τα συμβαλόμενα μέρη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εργαζόμαστε για την βιωσιμότητα της αλίας και την καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Πολλές φορές βέβαια δυστυχώς εντοπίζουμε και εκεί μία πρόοδο που είναι πολύ αργή. Όσον αφορά τώρα στην πρόσβαση Yeah. So, um, the, um, the, the, the close... Μάλιστα όσον αφορά την ε, ρήτρα για την πρόσβαση σε πόρους στα πλαίσια των FMOs. Θέλουμε να θίξουμε το ζήτημα αυτό και στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται. Δεν θέλουμε να λέμε ότι θα πρέπει να ισχύει αυτό μόνο για τους ε, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να το θίξουμε το ζήτημα αυτό, αποτελεί συστημικό ζήτημα και πρέπει να τεθεί στα πλαίσια των FMO. Η πρόσβαση στους ε, πόρους θα πρέπει να είναι γενικότερα διαθέσιμη ή θα πρέπει να υπάρχει ένα τέλος όσον αφορά τους πόρους αυτού, την, πρόσβαση αυτούς τους πόρους. Θέλουμε λοιπόν να γίνει μια γενικότερη συζήτηση στα, στο, και αυτή είναι η πρόθεσή μας να λάβει χώρα η συζήτηση αυτή. Τώρα, η πρόσβαση των πλειοκτητών στις διμερείς συμφωνίες, η συμμετοχή του στις διμερείς συμφωνίες. Ως προς αυτό, πρέπει να σας πω ότι κατά περίπτωση θα αξιολογηθεί η δυνατότητα αυτή. Οι πλειοκτήτες καταλαβαίνετε ότι αποτελούν μέρος της παραγωγικής δύναμης σε πολλές ε, περιοχές. Επομένως, στις περιοχές εκείνες προβλέπονται μεγαλύτερα επίπεδα λίας, μπορεί να προβλεφθεί και μια μεγαλύτερη συμμετοχή των ε, πλειοκτητών. Κατά περίπτωση πάντως θα διευθυνθεί το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα την ε, τεχνολογική συνεργασία, για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει διαφορά από την μία συμφωνία στην άλλη. Πρέπει να δούμε τι ανάγκε προκύπτουν κάθε φορά, ποιε είναι οι πραγματικές τεχνολογικές ανάγκες που έχουμε, ποιε είναι οι ανάγκες των κρατών, ποιε είναι οι, δυνατότητε απορρόφηση αυτή τη νέα τεχνολογία. αυτής επίσης. Αν δηλαδή μπορούν πραγματικά να εφαρμόσουν την συνεργασία αυτή στον τεχνολογικό τομέα. Θέλουμε να προωθήσουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την, το διαφορετικό τεχνολογικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η κάθε χώρα και όπου υπάρχει πιο έντονη αλλιευτική δραστηριότητα, τότε στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να προωθούμε τέτοια προγράμματα και να προβλέπουμε και την καλύτερη δυνατή διαχείριση των προγραμμάτων αυτών. Προγράμματα για την επιτήρηση των αλλιευμάτων και την εποπτεία που πρέπει να υπάρχει όσον αφορά τα αλληλευτικά αποθέματα. Επίσης θέλουμε να δούμε εκ νέου την τομεακή συνεργασία και θέλουμε να την κατευθύνουμε στον δρόμο του εξορθολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά στα οποία αναφέρθηκα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you, colleagues. Thank you. Ευχαριστώ Ευχαριστώ, ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ την Επιτροπή. Δεν έχω τη βεβαιότητα ότι ικανοποιήθηκαν με την απάντησή σας ε, οι συνάδελφοι κύριε της Επιτροπής, διότι υπάρχουν πολλά θέματα. Με τη σημείωση αυτών ε, τιμούμε ιδιαίτερα την παρέμβαση του συναδέλφου όσον αφορά τέτοιου είδους συμφωνίες. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε σε βάθος και να το εξετάσουμε σε βάθος. Κύριε Κατά, και εσείς νομίζω ε, κάνετε λόγο για τις προσωρινές συμφωνίες ε, ή και τη διακοπή τους. Είναι κάτι που συμμεριζόμαστε ως απογοήτευση του να υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες ε, και να εξετάζουμε εμείς αυτές τις συμφωνίες όταν πια έχουν αποφασιστεί από το Συμβούλιο, έχουν εγκριθεί και βρίσκονται και λειτουργούν εδώ και μήνες κιόλας. Είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε και να πούμε τι, ποιες είναι οι απόψεις μας ως Ευρωκοινοβούλιο για αυτά. Πρώτον δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με αυτή την κατάσταση. Και κύριε Μιλάνα κάνατε εσείς λόγο και αναφέρατε πολύ σκόπιμα ερωτήματα για το τι είναι αηφόρο. Τι είναι αηφόρες συμφωνίες αλληλείας. Εγώ θα το προσέγγιζα, υπάρχουν δύο τουλάχιστον πράγματα που πρέπει να εντάσσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Περιβαλλοντική αηφορία είναι το ένα και το άλλο είναι γενικότερη κοινωνική αηφορία ως θέμα. Αναφέρθηκαν οι προδιαγραφές του Διεθνούς Γραφείου, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τους ε, αλληλείς και πρέπει να δούμε σε σχέση με τις εταιρικές συμφωνίες αλληλείας και όσους απασχολούνται μέσα σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει ένα κενό κάποιο κενό για αυτά τα θέματα. Κάνουμε λόγο για προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας στις συμφωνίες και στα πρωτόκολλα και όλα αυτά, αλλά οι προδιαγραφές για τους αλληλείς του Διεθνού ε, Οργανισμού Αλίας και τους ε, εργαζόμενους στην Αλία δεν είναι εξειδικευμένε προδιαγραφές όπως εκείνες που ισχύουν για άλλα επαγγέλματα. Πρέπει να το δούμε από πλευρά ορισμού. Και αν θέλουμε να έχουμε ρήτρε ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες και για την ευδοκίμησή τους, πιστεύω ότι και οι Ευρωπαίοι πλειοκτήτες θα πρέπει να κάνουν την προσπάθεια να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στις ε, διατάξεις ε, για τους αλληλείς ε, του Διεθνούς Οργανισμού Αλληλείας και πρέπει αυτό να πιέσουμε να γίνει. Έτσι να μπορούν να λειτουργούν όλα αυτά υπό τις συμφωνίες για την αλληλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή ιδέα θα ήταν αυτό. Ευχαριστώ που αναφέρθηκε από όλους η καταπολέμηση της παράνομης και λαθρέας αλληλείας ως προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα. Η κυρία Φράγκα επίσης τόνισε κάτι τον ρόλο <clears throat> των περιφερειακών οργανώσεων αλληλείας και τον μη ικανοποιητικό τρόπο που ε, αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ε, συμβατικά, ε, συμβατικούς εταίρους. Είναι μεγάλη η πρόκληση ώστε να υπάρξει μεταρρύθμιση, ώστε να υπάρχουν κυρώσεις αυστηρές για εκείνους που δεν συμμορφώνονται. Για την πειρατεία, θέμα το οποίο ανέφερε η Πρόεδρος προηγούμενα. Η πειρατεία είναι πραγματικά ανησυχητικό παράγοντας και για να αποφύγουμε τέτοιες περιπτώσεις πειρατείας πρέπει να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο ότι θα λειτουργούμε με αηφόρο δίκαιο τρόπο όταν αλλιεύουμε σε χωρικά υδατά τρίτων χωρών. Με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα και να θεωρούν ε, οι τοπικοί πληθυσμοί ότι μέσα σε ένα πλαίσιο άδικο ε, διαδραματίζουμε εμείς ε, την, αναπτύσσουμε την αλλιευτική προσπάθεια. Υπάρχει μια τραγική κατάσταση και στην Σομαλία αλλά και για την Δυτική Αφρική κιόλας έχει αναφερθεί. Πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι στην ε, διεθνή, στην παγκόσμια σκηνή με υπεύθυνο τρόπο να δρούμε ώστε να αποφεύγουμε τέτοιες εκρήξεις βίας και πειρατείας. Η κυρία που ανέφερε τα ανθρώπινα δικαιώματα και που πρέπει να έχουμε καλό, λειτουργικού, καλούς λειτουργικούς ορισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω υπάρχει ένας τέτοιος ορισμός στη Συμφωνία Κοτονού, αλλά θα πρέπει να, το, να επαληθευτεί αυτό. Τώρα, για την τομεακή υποστήριξη ρώτησε η κυρία Φράγκα πώς μπορεί να δικαιολογηθεί το ότι 20 εκατομμύρια δίνονται στη Μαυριτανία και πολύ λιγότερα 2 εκατομμύρια στην Κινέα Μπισάου. Πρέπει να πούμε ότι ναι, αν θέλουμε να αποσυνδέσουμε τα δύο αυτά, θα πρέπει να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι ανάγκες των ε, ε, επιμέρους χωρών και πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις ε, Πολλά ενδιαφέροντα σχόλια λοιπόν και ερωτήσεις είχαμε και προσβλέπω στη συνέχεια των συζητήσεων και με τους κοιόδης και τους συγητές και την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Λεβίν. Κύριε Ντεπίπερ. Λοιπόν, για να δούμε με τη σειρά. Bueno, nada, Όχι, εντάξει, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτού του θέματος στις επόμενες συνεδριάσεις μας προβλέπεται καταρχήν από πλευρά χρονοδιαγράμματος ότι τον Απρίλιο θα ψηφιστεί προς έγκριση να έχουμε και αρκετές επιτροπές για την εξέταση αυτού του θέματος. Ολοκληρώνεται το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη και περνάμε στο επόμενο, στο 7 που είναι η κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα της αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Εισηγητής ο κύριος Στίβενσον. Θα εξετάσουμε ακριβώς αυτή την νομοθετική πτυχή, θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Τι θέλετε, να μιλήσετε πρώτα εσείς κύριε Στίβενσον ή η Επιτροπή. Εσείς ή επιτροπη εσεις η επιτροπη τι λέτε. Okay, yeah. Λοιπόν, ορίστε, έχετε τον λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. ήθελα να πω το Διαμόρφωσα αυτή την πρόταση σε 20 ερωτήσεις. Αυτός είναι ένας κανονισμός και εν τελική αναλύση θα πρέπει να θα υπάρξουν σε μια σειρά ολόκληρων τροπολογιών και καμία φιλτουμία. Προσπάθησα αυτή τη στιγμή να προλάβω να μην υπάρξουν πολλές τροπολογίες, διότι είναι ένα μίσο θέμα και βεβαίω είναι νομοθετικού περιεχομένου για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ευρεία. Σε αυτή τη φάση λοιπόν για να γίνει πλήρες και αντιληπτό ξεχώρισε αυτό σε 20 ερωτήσεις και επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή να περάσω σε αυτά τα θέματα με σύντομες απαντήσεις που θα δίνονται σε κάθε φάση. Και θα ήθελα να ακούσω βέβαια τις απόψεις επί αυτό το ερωτών. Πρώτον, θα πρέπει θα πρέπει τα οι οργανώσει χαλαριγών θα πρέπει να, πρέπει να παίζουν ένα ρόλο σημαντικό. Ναι, θα πρέπει να γίνει η απάντηση. Οι Βρυξέλλες θα πρέπει να, συζητεί, να θέτει το βασικό πλαίσιο όσον αφορά τις κοινή πολιτική ε, και η κράτη μέρα θα λαμβάνει την ευθύνη για την εφαρμογή τη, με τις παραγωγούς για την εξέλιξή της οι Βρυξέλλες θα πρέπει να δίνουν μια σειρά δυνατοτήτων επιλογών για να είναι κατάλληλες αυτές για την δική τους και βεβαίως θα πρέπει να σέβονται τη, τα τεχνικά θέματα καθώς επίσης και τις ποσοστώσεις. Αυτό το πρώτο. Δεύτερο, πώς θα αποφύγουμε πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη συγκέντρωση στα χέρια όλων σε πολυεθνικών Νομίζω πως την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την νομική επιτροπή που είπε την άποψή του για τις, παρα, για παραχωρήσεις που γίνονται όσον αφορά το θέμα αυτό, ότι είναι νόμιμες είπες, αλλά δεν μπορεί να οι μεταφορές να γίνονται με περιορισμούς. Εάν αν το TFC λοιπόν ε, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και όχι ε, Θα πρέπει αυτές οι συμφωνίες λοιπόν να γίνονται σε 15 ετή σειρά. Τρίτο, όσον αφορά τη δακολογία, τις υπερεθνικές παραγωγούς, τους τοπικούς παραγωγούς, θα πρέπει να υπάρχει μια σαφήνεια όσον αφορά αυτό στις οργανώσεις παραγωγών. Στην Ιρλανδία υπάρχουν τρεις μόνο. Υπάρχει, στην Ολλανδία υπάρχει μόνο στο Ιδρύμα Βασίλειο 26, στην, στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία και δέκα από αυτά είναι στην, στην ε, Σκοτία. Επίσης στην Γαλλίση υπάρχουν δέκα. Νομίζω πως οι μικρές λοιπόν παραγωγικές μονάδες θα πρέπει να είναι και οργανώσεις θα πρέπει να είναι ικανές να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα, τη δική τους βιωσιμότητα. Οι υπερεθνικές, οι διεθνείς ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται στη Μεσόγειο. Σε διάφορες χώρες ε, στην Ιρλανδία για παράδειγμα ε, ήταν το ιδεώδες μέρος για να δημιουργηθούν αυτές οι υπερεθνικές ή διεθνείς και για να μην υπάρχουν αυτές οι δεσμευτικές νομοθεσίες οι οποίες υπάρχουν. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια συγχώνευτη σε αυτό το ποιόν και όχι μια ε, συνεργασία μεταξύ τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ούσα μια ελεύθερη αγορά δεν θα πρέπει να θέτει ε, κανονισμούς από το κέντρο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία, αυτό που βλέπουμε μετά από πολλές συνεδρίες που γίνονται, και να υπάρχει ανοιχτή πάντως στον ανταγωνισμό. Πέμπτο, πέμπτο, μπορούν αυτές οι οργανώσεις να παίξουν το ρόλο που πρέπει να παίξουν. Σύμφωνα, το 23% είπε η Επίτροπος των αλλιευμάτων πέφτουν στο νερό, εξαφανάζουν. 7 εκατομμύρια τόνοι είναι αυτοί. Γιατί αυτά πέφτουν στο νερό, εξαφανίσουν, διότι είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα αλλιεύσης, να μην γίνονται αλλιεύματα τα οποία είναι παραλλιεύματα και τα οποία είναι άχρηστα έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο η ιερία θα γίνει και οικονομική αλλά και βιολογική και η Κομισιόν αυτή τη στιγμή ο μόνος σκοπός που θέτει είναι το βιολογικό. Χωρίς όμως μια βιωσιμότητα οικονομική τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολο και τη βιολογική βιωσιμότητα εφόσον θα πρέπει να υπάρχουν ε, κανόνες οι οποίες διέπουν αυτή την κατάσταση και ότι ε, οι παραγωγικές ομάδες θα πρέπει να ε, αφήνονται ελεύθερες να δράσουν όπως θέλουν. Έκτο θέμα, ερώτηση. Θα πρέπει, θα πρέπει αυτά τα αριώματα τα οποία σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να γίνουν στις επικυβερνητές οργανώσεις, ναι ή όχι. Εάν αυτά είναι Εάν αυτά τα πράγματα δοθούν σε μη κυβερνητικέ οργανώσει και φιλανθρωπικέ, θα είναι αυτό καταστροφικό. Δηλαδή, το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι, είναι να χρησιμοποιηθεί σαν ε, ηχθιόλαδο και βεβαίω με τις ατάλληλες επιδοτήσεις που πρέπει να δίνονται στον παραγωγό, στον αλλιέμπρο κειμένο υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί τεχνολογίες μέσα ηλεκτρονικής αγοράς στην ΕΕ με διάφορα συστήματα VMX και άλλα και κατά πόσο πραγματικά μπορούμε να έχουμε πλήρη γνώση πού έχουν, πώς έχουν και πώς έχουν αλληλευθεί, από πού έρχονται, πού ε, ε, αποβιβάζονται, σε ποιο ε, λιμάνι και ούτω καθεξής. Κατά πόσο λοιπόν πραγματικά μπορεί να υπάρχει μια κάρτα στην οποία είναι όλα εγγεγραμμένα αυτά και να υπάρχει ένα είδος κάρτας όπως είναι η πιστοτική και μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να εγγράφει και να γνωρίζει πραγματικά από που ήρθε όλα τα στοιχεία του αλλιεύματος. Και κατά αυτόν τον τρόπο ε, ξέρετε, μου δεδείχθη αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει, μου έγινε επίδειξη και μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό το σύστημα όλες οι δραστηριότητες αλίευσης που γίνεται. Είναι ένα πλήρες σύστημα αυτό το οποίο υπάρχει και νομίζω πραγματικά μπορεί να είναι ευεργετικό για τους πάντες. Πού μπορούν να συντονιστούν τα αλλιεύματα, οι ελεύσεις και η δατοκαλλιέργεια. Πώς μπορεί να γίνει καλύτερο συντονισμός. Πότε λοιπόν μπορούν να περιμένουν την αγορά να έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει περισσότερα είδη, ποια είναι τα δότερα είδη, κατά πόσον αυτή τη στιγμή η παραγωγή οι οποίοι υπάρχουν να υφίστανται εκείνες τις υποχρεώσεις που υπάρχουν και, τα, και πώς θα υπάρξει η μεγαλύτερη απόδοση. Πώς μπορεί να γίνει μια βελτιοποίηση ε, όλης αυτής της για να φτάσουμε στο βέλτιστο κύριο σημείο της αγοράς. Ξέρετε, υπήρξε ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε όσον από την παράβαση στην, στην αγορά. Μπορούν λοιπόν όλα αυτά να χρησιμοποιηθούν και μπορώ να πω με ε, ανάμεικτες απόψεις οι οποίες εκ μέρους των παραγωγών όπως υπήρξε μια συμφωνική συμφωνία και μερικοί είπαν ότι αυτή η δυνατότητα που δόθηκε προκάλεσε τις τιμές και υπήρξε ε, παρέμβαση με ελεύθερη, στην ελεύθερη αγορά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ότι στην ελεύθερη αγορά χρειάζεται μια παρέμβαση και είναι κάτι το οποίο άκουσα και στο Λονδίνο. Το καλύτερο, ε, είπε στο Λονδίνο, ε, η αποθήκευση είναι η, αγορά, η θάλασσα, συγγνώμη, η καλύτερη αποθήκη είναι. Έτσι λοιπόν, για να μην υπάρξει μεγάλη αποθήκευση, ποιος θα, όταν υπάρχει αποθήκευση, ποιος θα πληρώσει, πώς θα χρησιμοποιηθεί για εκείνα τα είδη όπως είναι οι μικροσαρδέλες, οι αντσούγες και ούτω καθεξή. Το ηχθιέλαιο. ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν ψηλές τιμές όλα αυτά, αλλά υπάρχει μια γενική άποψη ότι θα πρέπει να ε, χρησιμοποιείται η αποθήκευση όταν είναι αναγκαία να γίνει, διότι είναι πάρα πολύ ακριβή και εφόσον δεν υπάρχουν ψάρια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν αποβάλλονται και πόσο μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρξει μία πλήρη κάλυψη όλων αυτών με μία πολιτική η οποία θα σε αυτό το τομέα. Επίσης, υπήρχε διαδεδομένη άποψη ότι η Κομισιό ήταν αυτή που θα πρέπει να έχει εισάγει ένα κονισμό για μια ε, ετικέτα οικολογική eco-label και αυτό νομίζω αν γίνει αυτό θα μπορώ να γίνει πολύ πιο ευπρόσδεκτο με μέρους του κοινού. Ποια θα, τι θα πρέπει να συμβάνεται στην πληροφόρηση που θα πρέπει να γίνει με αυτό το eco-label προς τον κόσμο. Νομίζω πραγματικά ότι το κοινό θα ξέρει πάρα πολύ καλά πότε αλλιεύτηκε, αυτό θα είναι, δεν θα είναι υποχρεωτικό, αλλά πότε έχει αποβιβαστεί από το πλοίο και αυτό θα είναι που ζητάει ο καταναλωτής. Πιστεύω πραγματικά θα υπάρξουν με, με τις περιοχές αλλιεύσεις, πιστεύουμε πως πραγματικά κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφευθεί αυτό το που γίνονται με το παγόνο-ξεπαγόνο και θα υπάρξει μια ετικέτα η οποία θα είναι κοινή ε, ένας κοινό παρονομαστής ο οποίος θα λέει πραγματικά πότε συνελήφθη, πότε σκοτώθηκε και πότε μπήκε στο, στην κατάψυξη. Υπάρχει μία γενικότερη άποψη ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή ο κανονισμός που έχει εκτός ΕΟΚ θα πρέπει να υπήρχε και εντός ΕΕ. Θα πρέπει να υπάρχει χώρα παραγωγής, η χώρα καταγωγής και από που ε, όχι μόνο που έχει σφαγιαστεί, αλλά που έχει εξαχθεί μέχρι να φτάσει στα χέρια μας. Και τέλος, η, η ε, θα πρέπει να έχει το δικό της ποιοτικό έλεγχο ο οποίο θα, θα γίνεται για να δοθεί το eco-label, αυτό το οικολογικό, το οικολογικό συγγνώμη, ε, ετικέτα. Έτσι το κοινό θα χαιρετίζει και θα, ε, θα χαιρετήσει αλλά και θα υποδεχθεί αυτές τις προσπάθειες που θα γίνουν και αυτά τα ψάρια τα οποία θα έχουν αυτό το, ε, την ετικέτα. Νομίζω πως αυτό είναι σημαντικό και είναι απαραίτητο, να έχουμε στάνταρ οργανισμό, στάνταρ ε, μέγεθος ψαριών, νομίζω πως πραγματικά οι οικολογικές οργανώσεις δεν θα δεχθούν κάτι τέτοιο να γίνει. Τα μη μέλη ε, θα μπορούσαν να οδηγηθούν με το, χρόνο, με το ζόρι να συμμετέχουν. Νομίζω πως θα χρειαστεί να συμφωνήσουν, αλλά δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν με το ζόρι να κάνουν κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τα στάνταρ της αγοράς, τις προδιαγραφές, κατά δεν μπορούν τέτοιου είδους να εισαχθούν και κατά πόσο μπορούν αυτά να συνάδουν με τους προηγούμενους κανόνες κατά πόσο μπορούν να αληφθούν ευθύνε για αυτά τα θέματα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Κομισιόν και πώς αυτή η εφαρμογή θα γίνει. Η εφαρμογή βέβαια άπτεται στους παραγωγούς και μόνο και η κοινότητα μπορεί απλούστατα να βάλει το ελάχιστο μέγεθος το οποίο πρέπει να έχουν και μερικά ήδη θα πρέπει να λάβουν την επιστημονική γνωμοδότηση που χρειάζεται για την αλίευσή τους. Οι προτάσεις αυτή τη στιγμή της Κομισιόν όσον αφορά τη συλλογή καθώς επίσης και την κατανόηση αυτή που θα πρέπει να γίνει των πρακτικών υπάρχει μια γενικότερη συνένεση ότι η πληροφόρηση που θα πρέπει να έρχεται εκτό της αγοράς θα πρέπει να βελτιωθεί, θα πρέπει να υπάρχει πληροφοριοποίηση όλων αυτών όσον αφορά την αποβίβαση, τη μεταφορά πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και πώς πραγματικά να πρέπει να ληφθούν και περιβαλλοντολογικά θέματα υπόψη. Ένα σύστημα δηλαδή το οποίο θα μπορεί να μας λέει ότι online πόσο, πόσο η ρόγκα έχει αποβιβαστεί χθε, για παράδειγμα και που βρίσκεται και ούτω καθεξή. Τι ρόλο μπορούν να παίξουν αυτή τη στιγμή οι συνολικές αλληλευτικές επιχειρήσεις χρειάζεται περισσότερο να Ξέρετε ότι υπάρχει όλο και περισσότερη ζήτηση των αλλιευμάτων. Βεβαίω, οι υδατοκαλλιέργειε θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο και αυτή η οργάνωση η οποία υπάρχει δεν έχουν προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν για την υδατοκαλλιεργία. Θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη και ξέρετε, σε όσον αφορά την υδροτοπαλλεργία υπάρχουν αυτή τη στιγμή περί μεγάλη υποστήριξη για την ύπαρξη αυτών των κανονισμών και ιδιαίτερα για τη δράση την οποία θα μπορούν να αναπτύξουν σε αυτό το τομέα. Θα μπορούσε Όσον αφορά το Ταμείο για την Αλία, μπορούμε να δώσουμε το ποσό των 6,5 δισεκατομμυρίων όταν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες ακόμα και όταν δεν υπάρχει απαραίτητη διαφάνεια. Και τέλος, συμφωνείτε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την χρήση πράξεων κατά εξοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να υπάρχει το απαραίτητο επίπεδο ευελιξίας προκειμένου να μπορούν οι οργανώσεις παραγωγών να προσαρμόζονται στις αλλαγές οι οποίες αλλάζουν συνεχώς. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Αυτές πιστεύω ότι είναι οι βασικές ερωτήσεις, στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στην τελική έκθεση. Βέβαια, στην αδελφή μου μπορεί να έχουμε άλλες ερωτήσεις και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα τις ακούσω και θα ήθελα να ακούσω βέβαια και τις απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στις ερωτήσεις που ήδη ακούσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στρούαν Στίβενσον για την εργασία του, καθώς επίσης και για τις απαντήσεις που έδωσε στις 20 ερωτήσεις που θέτει. Είναι πολύ καλό, θέτεις και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, προφανώς και εμείς πρέπει όμως να απαντήσουμε περαιτέρω στις ερωτήσεις αυτές. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουμε προφανώς να προωθήσουμε την βιώσιμη αλία, να βελτιώσουμε την παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια αγορά, να βελτιώσουμε την ε, σύνδεση ανάμεσα στους παραγωγούς της αγοράς και την απόδοση της αγοράς αυτής. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε τις δυνατότητες κερδοφορίας προώθησης των ευρωπαϊκών προϊόντων, να υπάρχει ένα οικολογικό σήμα, όπως είπατε, να μειωθεί το διοικητικό άχθος. Αυτές είναι οι ευχές, τέλος πάντων, τις οποίες εμείς προωθούμε και συμφωνούμε βέβαια με τις προτάσεις που κάνετε κι εσείς. Ένα πρώτο ερώτημα. Όσον αφορά τα συλλογικά ταμεία προώθησης των αλληλευτικών προϊόντων. Δεν ξέρω ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα θέλει ουσιαστικά να πετύχει μέσω της πρότασης αυτής. Πρόταση η οποία βέβαια θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί, επομένως πρέπει να ξέρουμε πώς θα χρηματοδοτηθεί. Όσον αφορά τώρα τον μηχανισμό για την αποθήκευση, και το ζήτημα αυτό είναι ενδιαφέρον. Έχουμε, είναι ο μόνος μηχανισμός ρύθμισης αγοράς που απομένει στην πρόταση αυτή και πρέπει να έχουμε τη ρύθμιση των αγορών και χρειαζόμαστε ρύθμιση και για τα προϊόντα λίας και υδατοκαλλιέργειας. Το σύστημα μηχανισμού αποθήκευσης ε, επιτρέπει την αγορά προϊόντων από τους φορείς όταν η τιμή των προϊόντων αυτών ε, ε, κατεβαίνει κάτω από την, αποφασισμένη τιμή. Μπορούν λοιπόν να αποθηκευτούν τα προϊόντα αυτά και στη συνέχεια να διατεθούν στην αγορά αυτός ένας κανόνας που υφίσταται στην αγορά και μπορεί να συνεχίσει να ισχύει. Αποφεύγεται κατά αυτόν τον τρόπο η διανομή των προϊόντων, κάτι το οποίο δεν είναι ευκταίο και επίσης αποφεύγεται και η καταστροφή των προϊόντων και εξισορροπείται καλύτερη αγορά κατά αυτόν τον τρόπο. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να αποθηκεύουν τα προϊόντα. Πρέπει να γνωρίζουμε γιατί αποθήκευση μιλάμε. Στρού, αν αναφέρθηκε σε αυτό, θα προβλέπονται κάποια συστήματα κατάψυξη και πώ θα γίνεται αυτό το πράγμα. Πόσο χρόνο μπορούμε να διατηρήσουμε τα προϊόντα αυτά. Και δεν θα πρέπει η τιμή εκκίνησης να τίθεται σε τέτοιο επίπεδο που να τελικά προωθεί περισσότερο να ευνοεί την αποθήκευση των προϊόντων και όχι την πώλησή τους. Ο μηχανισμός λοιπόν αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται από μια ξεκάθαρη χρηματοδότηση και ο μηχανισμός αυτός λοιπόν θα πρέπει να χρηματοδοτείται, να χρηματοδοτείται με συγχωρείτε, με τρόπο ευφυή και αηφόρο. Όσον αφορά το οικολογικό σήμα τώρα, προφανώς είμαι υπέρ του να αρχίσει να χρησιμοποιείται ένα ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Βέβαια υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στην προτινόμενη κοινή οργάνωση αγοράς που έχει ως στόχο να ενημερώνει καλύτερα τον καταναλωτή και την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμεί να πετύχει μια εναρμόνιση μέσω της θέσπισης αυτής της κοινή οργάνωσης αγοράς. Και τίθεται ένα ερώτημα. Θέλουμε να διατηρήσουμε το σύστημα εξαιρέσεων παρεκκλήσεων όσον αφορά την χώρα προέλευσης, όπως έχουμε με την Γουινέα Μπισάου και που επηρεάζει συμφωνίες που έχουμε για διάφορα είδη όπως ο τόνος. Υπάρχει μία αντίφαση ως προς τους στόχους που παραθέτουμε στην πρόταση αυτή και αυτά τα οποία ισχύουν στην πράξη. Είναι πολύ σημαντική πάντω η εργασία που έκανε Στρούαν, το ότι καταφέρνει και βελτιώνει την αρχική πρόταση για τη δημιουργία αυτή τη κοινή οργάνωση αγορά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ Στρούαν για την διεξοδική αυτή εργασία σου, για αυτό το πλήρε έγγραφο εργασία. Πραγματικά κατάφερε να καλύψει πάρα πολλά πράγματα και απορώ πως η γραμματεία σου επέτρεψε να γεμίσει τόσε πολλέ σελίδε, 14 συνολικά. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις ερωτήσεις τις οποίες θίγεις, θα κάνω κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις για συγκεκριμένα σημεία. Ο γενικότερος ε, στόχος της νέας κοινή οργάνωσης αγοράς είναι να επιτρέψουμε τελικά στους ε, αλείς να έχουν καλύτερες αποδοχές στα πλαίσια μιας πιο βιώσιμης ε, αλίας. Θέλουμε ουσιαστικά να προσδώσουμε μια προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους, να και το να δυναμώσουμε τις οργανώσεις παραγωγών νομίζω ότι αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και συμφωνώ και με την πρότασή σου να συγχωνευτούν οι οργανώσεις παραγωγών προκειμένου να γίνουν πιο ισχυρές απέναντι στους λιανοπολιτές. Έχουμε δει ότι υπάρχει ένα ολιγοπόλιο όσον αφορά τη θέσπιση των τιμών και υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στις αποδοχές των των αλλιευτών, την τιμή που θέτουν για τα προϊόντα τους και την τιμή που τελικά πληρώνει ο καταναλωτής για τα προϊόντα αυτά στην αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η συγχώνευση των οργανώσεων παραγωγών ουσιαστικά θα ενδυναμώσει και την θέση τους. Επίσης, αναφέρεσαι στην υφιστάμενη CMO, την υφιστάμενη οργάνωση αγοράς, όπου υπάρχει ένα κεφάλαιο για το εμπόριο, το οποίο δεν υπάρχει στη νέα πρόταση. Αυτή είναι μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποιο λόγο δεν βλέπουμε πλέον αυτό το κεφάλαιο. Επίσης, αναφέρθηκες πολύ στις απορρίψεις. Μια ερώτηση έχω για εσένα, Στρούαν. Είπες ότι μίλησες με πολλούς παράγοντες της αγοράς. με πόσους τελικά μίλησες και τι είδους παράγοντες της αγοράς ήταν αυτοί όταν μας λες ότι σου δώσαν όλες αυτές τις απαντήσεις τις οποίες παραθέτεις. Όσον αφορά πάντως τις απορρίψεις, τα απορριπτόμενα λιεύματα, ανησυχώ ιδιαίτερα κάθε φορά που βλέπω ότι ε, οι οργανώσεις παραγωγών θέλουν επιπλέον 23% στις ποσοστώσεις. Γιατί τόσο είναι και το ποσοστό τελικά των απορριπτώμενων αλλιευμάτων. Στόχος μας δεν είναι να συνεχίσουμε να αλλιεύουμε τόσα πολλά ψάρια προκειμένου να προχωρούμε και σε τόσο μεγάλες απορρίψεις. Στόχος είναι να παραμείνουν τα αλλιεύματα αυτά τα οποία δεν επιθυμούμε να αλλιεύσουμε στο νερό, μέσα στη θάλασσα. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να δοθούν οι πόροι αυτοί προκειμένου να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το φαινόμενο της παρεμπίπτους ασαλίας. Θα μπορούσαμε πάντως να υποστηρίξουμε την όλη προσπάθεια προκειμένου να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση των ε, αλλιευμάτων εκείνων που ε, κατά λάθο ουσιαστικά αλλιεύονται και στη συνέχεια εκφορτώνονται και απορρίπτονται. Θα μπορούσε αυτό να μα βοηθήσει, να βοηθήσει του επιστήμονε τουλάχιστον να κάνουν καλύτερε εκτιμήσει όσον αφορά του λευτικούς πόρου, δηλαδή τι αλλιεύεται από τη θάλασσα και τι καταλήγει στην απόρριψη μετά. Να σας πω και το νορβηγικό σύστημα το οποίο έχουμε, ένα 25% της, αξίας, της, της εμπορικής αξίας των αλλιευμάτων πηγαίνει στον ψαρά, και αν μπορεί να προωθηθεί στην αγορά στη συνέχεια πωλείται ως ε, αλλιευτικό προϊόν και τα έσοδα από τις πωλήσει αυτές ε, επιστρέφουν στο όλο σύστημα. Επομένως, ε, ο έλεγχος αυτός χρηματοδοτείται εν μέρη από τα χρήματα αυτά. Θεωρώ ότι το σύστημα είναι πολύ καλό, λειτουργεί πολύ καλά στην Νορβηγία. Το ερώτημα που θέτω λοιπόν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι για ποιο λόγο δεν προτείνει το σύστημα αυτό στην πρότασή τη. Όσον αφορά του φιλανθρωπικού οργανισμού, συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Δηλαδή υπονομεύει ουσιαστικά την αγορά το να δίνουμε δωρεάν ψάρια κατά αυτόν τον τρόπο. Εν γέννη θα πρέπει να αποφεύγουμε να αλλιεύονται τα ψάρια αυτά, ας μην δικαιολογούμε την αλλίευσή τους, λέγοντας ότι μπορούμε να τα δώσουμε στους φτωχούς στη συνέχεια, να, κάνουμε, να δημιουργήσουμε βιοκαύσιμα ή καλλιντικά. Ας λέμε εξ αρχής ότι αυτά τα ψάρια δεν έπρεπε να είχαν αλλιευτεί κάτι πολύ ενδιαφέρον, market intelligence, περισσότερες πληροφορίες στα πλαίσια της αγοράς, πώς μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να βλέπουμε τι γίνεται στις θάλασσες, πώς εξελίσσεται η ελευτική δραστηριότητα, πολύ θετική παρατήρηση σου αυτή, γιατί έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία προκειμένου να μπορούμε, προκειμένου να, μπορούμε να επιτηρούμε παντού τι γίνεται. Επομένως, το επιχείρημα που χρησιμοποιείς θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα βάσιμο και θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και στα πλαίσια του οικολογικού σήματος και της ιχνηλασιμότητας. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι αλλιεύεται, πού αλλιεύεται, ποια χρονική στιγμή, ποιο είναι το είδος το οποίο αλλιεύεται και τι αλλιευτικό εργαλείο χρησιμοποιείται για την αλλιεύση του συγκεκριμένου αλλιεύματος. Αυτή την πληροφορία ακριβώς χρειάζονται οι καταναλωτές. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε για να έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία. Συζήτησα το ζήτημα αυτό με εκπροσώπους ορισμένων κρατών μελών και μου είπαν ότι με αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια υπερβολική επιτήρηση εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και ότι στην πράξη μπορούσε να μην υλοποιηθεί. Αλλά νομίζω ότι σε συνδυασμό με τις απαγορεύσεις για τις απορρίψεις, σε συνδυασμό με όλους τους κανονισμούς που έχουμε για την επιτήρηση, μπορούμε να προβλέψουμε μια τέτοια εποπτεία. Για ποιο λόγο να μην έχουμε την εποπτεία αυτή και για την αλλιευτική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο να μην έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες για το καταναλωτή. Τι αλλιεύεται, πού αλλιεύεται και ποιο έχει αλλιεύσει το συγκεκριμένο προϊόν. Για το κρέας, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ακριβώς από ποιο αγρόκτημα προέρχεται το βοδινό ή το πουλερικό το οποίο αγοράζει ο καταναλωτής. Οι καταναλωτέ χρειάζονται τι πληροφορίε αυτέ, επομένω νομίζω ότι και στον ηλεκτρικό τομέα θα πρέπει να τι έχουμε. Όσον αφορά το οικολογικό σήμα και ολοκληρώνω με αυτό, δεν είμαστε ιδιαίτερα υπέρ ενό ευρωπαϊκού οικολογικού σήματο. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει κάποια κριτήρια για το τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε ένα τέτοιο οικολογικό σήμα, δηλαδή κάποια ελάχιστα κριτήρια, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει το δικό τη το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα. Α θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ αυστηρά περιβαλλοντικά στάνταρτ για όλου, πρότυπα, με συγχωρείτε, για όλου του αλληλεί αλλά δεν νομίζω ότι είναι ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει ένα ενιαίο και μοναδικό ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα. Και όσον αφορά την ερώτηση παριθμών 13, νομίζω ότι στην ερώτηση αυτή συναντούνται οι δύο εκθέσεις μας, όσον αφορά δηλαδή το ισότιμο αυτό επίπεδο ανταγωνισμού ανάμεσα στα προϊόντα των δικών μας των αλλιέων, καθώς επίσης και τα προϊόντα αυτά τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες. Εδώ βρίσκεται το βασικό ζήτημα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό και μπορούμε να θέσουμε στις εισαγωγές περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Θα εμποδίσει με τέτοια, προτεθή, μια τέτοια πρόθεσή μας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, θα εμποδίσει με τέτοια πρόθεσή μας ακόμα και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν θέλουμε πάντως σήμερα να είμαστε πραγματικά υπεύθυνοι, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις εισαγωγές τα συμφέροντα των ε, Ευρωπαίων αλλιέων, καθώς επίσης και όσων ασχολούνται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, συγκλίνουν στο σημείο αυτό. Θέτω λοιπόν το ερώτημα αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα απαντήσετε εσείς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ερώτηση 13 του Στρούαν Στίβενσον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την δουλειά που κάνατε, που είναι σημαντική υπόθεση. Σύντομα, όπως ε, και σύντομα αναφέρθηκα στην προηγούμενη παρέμβασή μου, από πλευράς ουσίας η Ζάμπερ έχει δίκιο. Έχει δίκιο όταν λέει ότι εδώ έχουμε ένα από τα έγγραφα που πρέπει να διασφαλίζουν καλύτερο και περισσότερο εισόδημα για τους αλείς. Ταυτόχρονα όμως από την άλλη πλευρά αυτό θα πρέπει να προαγάγει και τα δικαιώματα των καταναλωτών και να έχουν εχέγγυα και να κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους οι καταναλωτές. Και εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο επί μακρόν έχουμε συζητήσει. Ουσιαστικά το γεγονός ότι έχουμε απουσία ευρωπαϊκής παραγωγής ή η ευρωπαϊκή παραγωγή φθήνει, συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Χάσαμε μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια αηφόρο υδατοκαλλιέργεια ως τομέα κατά τα τελευταία χρόνια. Και βλέπουμε όλο και περισσότερο εισαγωγές ηχθείων και αποθεμάτων ηχθιακών από άλλες χώρες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει σίγουρα να λάβουμε υπόψη και να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών συνολικά, σφαιρικότερα, βλέπουμε ότι πρέπει να αναφέρουμε όλες τις παρατηρήσεις μας τώρα για τα σήματα labeling και την υδατοκαλλιέργεια ε, aquaculture, labeling and aquaculture. Νομίζω όμως κάποια σχόλια θα έπρεπε γενικότερα να γίνουν. Δηλαδή, μεταξύ αυτών πρώτα απ' όλα, το ότι δεν έχουμε αναπτύξει την υδατοκαλλιέργεια επαρκώς ικανοποιητικά ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μας. Χαμηλότερα δηλαδή επίπεδα παραγωγής ή α, ε, ηχθιακής παραγωγής. Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας τι σημαίνει. Σημαίνει ότι χρειάζεται σχεδιασμός, χρειάζεται ένας προγραμματισμός. Με άλλα λόγια, πρέπει να καθορίσουμε και να θεσπίσουμε όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίους λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά το εγχείρημα της υδατοκαλλιέργειας. Δηλαδή και οι δύο κανονισμοί, και αυτός και ο προηγούμενος που ήταν και είχαμε υποσυζήτηση, πρέπει να προβλέπουν στοιχεία που θα διασφαλίζουν ότι η θάλασσα, το υδάτινο περιβάλλον θα αποτελεί και για τις υδατοκαλλιέργειες ένα αποτελεσματικό, μια αποτελεσματική παράμετρο. Μία αναγκαία προϋπόθεση θα είναι η μεταρρύθμιση να συνεχίσει να συνεχιστεί και να αναπτύξει μια πολιτική αυτή η αναθεώρηση όπου τα αλλιεύματα, οι αλλιείς, οι αγορές, οι ποσοστώσεις, ο εξοπλισμός, όλα αυτά θα είναι η ή λύθη μιας ε, σφαιρικότερης ε, συνολικής πολιτικής που θα αναπτύξουμε. Δηλαδή, ο υδάτινος χώρος ε, ως τομέας, ως παράγοντας, σε κανένα από τα έγγραφα δεν αναφέρεται ούτε μια λέξη για τη θάλασσα και το υδάτινο περιβάλλον. Θα πρέπει έτσι να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την ιδέα για την υδατοκαλλιέργεια. Να προγραμματίσουμε και να σχεδιάσουμε συγκεκριμένους τομείς ως ε, λιθαράκια που θα συνθέτουν ένα πανόραμα, ένα μοσαϊκό. Εκ με όλες τις άλλες προσπάθειές μας. Πρέπει να εισαγάγουμε λοιπόν την ιδέα και να θεσπίσουμε την ιδέα, να την κατοχυρώσουμε ότι η θάλασσα, ο, ο υδάτινος χώρος, το υδάτινο περιβάλλον είναι το πλαίσιο όλων αυτών των δράσεων. Δηλαδή, η θάλασσα, το υδάτινο περιβάλλον και η αλληλεία και η υδατοκαλλιέργεια. Είναι θεμελιώδου σημασία αυτό. Αν θέλουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία συσχετίζονται και αλληλοσυνδέονται για τις επιπτώσεις των δράσεών μας να εξεταστούν σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την υδατοκαλλιέργεια. Ακούμε για την υδατοκαλλιέργεια ως μια στρατηγική, αλλά δεν υπάρχει input, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα και δράσεις ώστε να θεσπιστούν στόχοι και ε, σκοπή για την υδατοκαλλιέργεια. Δηλαδή να μην ε, βρισκόμαστε σε μηδενικό σημείο όταν κάνουμε λόγο για το, τις υδατοκαλλιέργειες. Από το 2009 μέχρι σήμερα δεν αναπτύχθηκε η υδατοκαλλιέργεια με κανένα τρόπο. Δεν προχωρήσαμε, δεν σημειώθηκε πρόοδος. Χρειάζονται λοιπόν εξειδικευμένες πληροφορίες να εξειδικεύσουμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε και θα πορευθούμε. Πρέπει να δούμε πώς μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί οι κλάδοι της ευρωπαϊκής παραγωγής όσον αφορά συγκεκριμένα την υδατοκαλλιέργεια στην παγκόσμια σκηνή, στην παγκόσμια αγορά. Χρειαζόμαστε μια βίο υδατοκαλλιέργεια, μια αηφόρο υδατοκαλλιέργεια που θα λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους του περιβάλλοντος και θα είναι αηφόρο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υποστηρίζεται μια τέτοιου είδου υδατοκαλλιέργεια. Προγραμματισμό και σχεδιασμό λοιπόν για τι ε, θαλάσσιε ε, δράσει και δραστηριότητε. Υποστηρικτικό πλαίσιο για αναπτυξιακέ πολιτικέ Αυτές οι ιδέες δεν θέλουμε να ενταλθούν, να αποσταλούν σε κάποιο άλλο πλαίσιο ή σε κάποιους άλλους αποδέκτες. Θα πρέπει να δούμε τις στρατηγικές γραμμές και δεσμευτικές δράσεις για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην υδατοκαλλιέργεια. Και μέχρι το, μέχρι το 2013 λέγεται πρέπει να αναπτυχθούν αυτές. Όμως δεν είναι δεσμευτικές. Και τέτοιου είδους αποδυναμωμένες δράσεις όπως μη δεσμευτικές δράσεις θα συνεχίσουν να οδηγούν η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την υδατοκαλλιέργεια σε ένα μικρό τομέα, ενώ έχει μεγάλο μείζωνα ρόλο να διαδραματίσει για την αύξηση της παραγωγικότητας. Και ένα τελικό σχόλιο εφόλων αυτών. Και συνδέω τα θέματα απόρριψης ηχθείων τώρα και μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Έχω αρκετά ερωτήματα για την ε, εκφόρτωση και την ε, εκφόρτωση ε, όσον αφορά ε, οι ηχθείες που, που θα έπρεπε να απορρίπτονται. Πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να δούμε αν είναι δυνατόν να παράγεται ηχθιέλαιο, ηχθιέλαιο ή αν είναι δυνατόν να έχουμε κάποια υποπροϊόντα από αυτά. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο σε τέτοια κλίμακα θα είναι ένα κίνητρο που θα δοθεί για την εκφόρτωση περαιτέρω τέτοιων παράλληλων αλλιευμάτων. Και υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους τέτοια παράλληλα ή παράπλευρα τέτοια αλλιεύματα μπορεί να βρίσκονται σε ένα σκάφος. Δεν πρέπει λοιπόν να πάρει διαστάσεις όλο αυτό. Όμως από την άλλη πλευρά, αν θέλουμε να εισαγάγουμε ένα στοιχείο το οποίο τα παράπλευρα αλλιεύματα θα τα οδηγεί στην επεξεργασία, στην ε, ηχθειοβιομηχανία, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι πόροι αλλιεύματα θα ε, συλλαμβάνονται, θα αλλιεύονται για την παραγωγή ηχθιελαίων, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην στρεβλώσουμε τα πλαίσια. Δεν γνώριζα για το, την νορβηγική αυτή εμπειρία ε, όμως ε, τα παράπλευρα αλλιεύματα είναι ένα ουσιώδες ζήτημα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν θεσπίζουμε και συν, ε, καταρτίζουμε κανόνες. Δεν θέλουμε οι κανόνες αυτοί να υπονομεύουν και να αποδυναμώνουν τον τομέα. Και δεν θέλουμε να αποδυναμώσουν και να οδηγήσουν σε ζημιές τους αλληλείς. Και μια τελευταία παρατήρηση για τα σήματα, labeling. Εδώ σε σχέση με τα όσα είπε η Ιζαμπέλ, σε άλλους τομείς στην Ευρώπη έχει θεσπιστεί μια πολιτική. Υπήρξε και μια έκθεση του Κοινοβουλίου που αφορούσε και, ε, ε, αναφερόταν στα θέματα made in ε, Italy, made in France, αλλά ως σήμα made in Europe, δηλαδή ευρωπαϊκό προϊόν. Να μπορούμε να πούμε ότι αυτού του είδους τα προϊόντα θα είναι προϊόντα ευρωπαϊκά που θα έχουν ουσιοδέστατο ρόλο να διαδραματίσουν στην παραγωγική αλυσίδα, διότι θα τα υποπτεύουμε αποτελεσματικά, δίνουμε ουσιοδέστατο ε, ρόλο και θέση, ουσιώδη θέση στην ε, διαδικασία εποπτείας και επόπτευσης. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μπορεί να συνεισφέρει ώστε η υδατοκαλλιέργεια να είναι βιώσιμη και αποτελεσματική. Διότι πρέπει να διασφαλιστεί, για παράδειγμα όταν έχουμε μύδια και ε, διάφορα από την Ιταλία ή η Γαλλία που δεν ε, ε, ανταγωνίζονται το ένα είδος το άλλο ή όταν έχουμε τέτοιου είδους προϊόντα όσον αφορά την ε, Ελλάδα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά υπάρχει πλεονέκτημα, πρέπει να υπάρχει πλεονέκτημα έναντι των προϊόντων που προέρχονται από την Ασία χωρίς όρους και προδιαγραφές και χωρίς σήμα ειδικών απαιτήσεων. Χρειάζεται λοιπόν ευρωπαϊκή σήμανση, ευρωπαϊκή ετικετοποίηση και ένα σήμα ευρωπαϊκό για να είμαστε αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί και να είναι κάτι το οποίο θα μπορούν να ταυτοποιούν και να αναγνωρίζουν με αυτό το ευρωπαϊκό προϊόν οι καταναλωτές. Αυτό πάλι με τη σειρά του θα σημαίνει ότι θα μπορούμε να ξεπεράσουμε την έλλειψη ε, ανταγωνιστικότητας στις τιμές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέιβις παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο οικολογικό σήμα. Ο Στρον Στίβενσον, πολύ σωστά στην έκθεσή του, αναφέρεται σε διάφορα ενδιαφέροντα ζητήματα σε σχέση με το οικολογικό σήμα. Μας λέει ότι ορισμένες οργανώσεις παραγωγών δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να πληρώσουν μια ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να τους δώσει ένα οικολογικό σήμα για την βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους, μα πρέπει να το κάνουν αυτό γιατί το ζητούν οι καταναλωτές. Στην έκθεση γίνεται μια φορά στην Βρετανία, αλλά νομίζω ότι είναι η Γερμανία αυτή η οποία χρησιμοποιεί ένα σύστημα πιστοποίησης περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος οργανισμός σούπερ μάρκετ, ένας πολύ μεγάλος όμιλος σούπερ μάρκετ στη χώρα αυτή που λέει ότι θα δεχθεί αλλιεύματα τα οποία φέρουν μόνο την οικολογική αυτή πιστοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό όταν παράγουμε κάτι, όταν πουλάμε κάτι προς τον καταναλωτή, προς τον πελάτη, να συμμορφωνόμαστε και προς πληροφορίες που θέλει το καταναλωτή. Ο Στρίουαν Στίβενσον επίσης μας λέει Προτείνεται μάλλον ότι θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία στο σύστημα, προκειμένου να υπάρχουν πολλά διαφορετικά οικολογικά σήματα τα οποία θα μπορέσουν να ισχύουν. Οτιδήποτε πρέπει να λειτουργήσει υπέρ του αλλιέως και υπέρ του, καταναλωτή, του πολιτή. Μα δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή μόνο για ένα τέχνασμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ενδεχομένω από του εμπόρους και του πολιτέ. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένε εγγύσει, γιατί διαφορετικά το όλο σύστημα θα είναι εντελώς αναξιόπιστο. Και ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά οικολογικά σήματα τα οποία υπάρχουν ε, και ισχύουν στην αγορά. Και ορισμένα από αυτά έχουν ε, επικριθεί. Πριν από 12 χρόνια, όταν ήρθα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, μιλούσαμε τότε για ένα eco-label, για ένα οικολογικό σήμα, το οποίο δεν πρόοδευε πάρα πολύ καλά και 12 χρόνια αργότερα δεν έχει ακολουθήσει πολύ θετική πορεία. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να θεσπίσουν ένα ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, τότε ουσιαστικά θα προσελκύσουν επικρίσεις από παντού. Οπουδήποτε ένα σκάφος κάνει κάτι το παράνομο, και εφόσον το σκάφος αυτό στη συνέχεια στα εμπορεύματά του χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα, τότε καταλαβαίνετε ότι το οικολογικό αυτό σήμα στη συνέχεια θα χάσει την αξιοπιστία του. κανεί, δεν θα το εμπιστεύεται πλέον. Α είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν με αυτό. Α εξετάσουμε όλα τα διαφορετικά οικολογικά σήματα τα οποία ήδη υπάρχουν στην αγορά. α εξολογήσουμε καταρχά πώ λειτουργούν τα σήματα αυτά και το να προσπαθήσουμε εμείς απλώς να δημιουργήσουμε το δικό μας το σήμα, τότε αυτό θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί θα προσελκύσουμε όλο και περισσότερες ε, επικρίσεις. Ο κύριος Γκάλαχερ έχει το λόγο. Uh, you, uh, First... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα με την πρώτη ματιά που ρίχνω στο έγγραφο αυτό να συγχαρώ τον Στρουασιμβέτσο να αποτελεί μια πολύ καλή βάση εργασίας και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις οι οποίες είναι πολύ θετικές, πολύ επικοδομητικές. Όσον αφορά το ρόλο των οργανώσεων παραγωγών, νομίζω ότι θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των αλλιευμάτων. Θα τον οπτύξω αυτό λίγο αργότερα. Σε ορισμένε χώρε υπάρχουν πολλέ οργανώσει παραγωγών. Στι περιπτώσει αυτέ θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμό των οργανώσεων παραγωγών. Σε κάποιε ε, χώρες από τρεις θα μπορούσαν να περάσουν σε δύο, σε άλλες μικρές χώρες η κατάσταση είναι πιο διαχειρίσιμη. Αλλά σε ορισμένες μεγάλες χώρες, όπως στην Ισπανία για παράδειγμα, έχουμε εκατοντάδες οργανώσεις παραγωγών. Νομίζω ότι θα πρέπει σε κάθε περιφέρεια να υπάρχουν τουλάχιστον, μάλλον να υπάρχουν το πολύ μία ή δύο οργανώσεις παραγωγών. Μπορούμε να μειώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την γραφειοκρατία, μπορούμε να εργαστούμε καλύτερα και θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί εν γέννη. Πιστεύω ότι ε, οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει σαφώς να συμμετέχουν στο όλο σύστημα. Όσον αφορά τις ε, συνολικές ελευτικές παραχωρήσεις, παράδειγμα από τη δική μου χώρα μπορώ να δώσω μόνο, νομίζω ότι το σύστημα αυτό αν συνεχίσει να ισχύει, θα ζημιώσει πάρα πολύ τον αλληλευτικό μας κλάδο. Οι αλληλευτικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιφέρειες της χώρας μου που δεν υπάρχουν άλλες οικονομικές δυνατότητες και τα μικρά σκάφη δραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι τα σκάφη αυτά τα οποία μπορούν να πάνε συγκεκριμένε περιοχές και μπορούν να επιστρέψουν στη συνέχεια σε κάποιους μικρούς λιμένες. Καταλαβαίνετε ότι ε, η κατάσταση δεν είναι η ίδια με τα μεγάλα σκάφη, τα οποία μπορούν να αλλιεύουν σε πάρα πολλές διαφορετικές περιοχές και μπορούν προφανώς να πηγαίνουν και σε όλους τους μεγάλους λιμένες. Το σύστημα συνολικών ελευτικών παραχωρήσεων πάντως θα πρέπει να είναι εθελούσιο και όχι υποχρεωτικό. Τώρα για τους αλείς. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν κάποια δικαιώματα διοκτησίας. Τα λιεύματα που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφά που ανήκουν στα κράτη-μέλη ανήκουν στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο αποφασίζει μέσω του συστήματος ποσοστώσεων ποιο έχει πρόσβαση σε τι. Και αν δεν υπάρχει βέβαια απαραίτητη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς και με του απαραίτητου κανόνε, τότε προβλέπονται και ε, κυρώσεις. Όσον αφορά τώρα το ρόλο που μπορούν να δραματίσουν οι οργανώσεις παραγωγών, μα μπορούν να δραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Από την 1η Ιανουαρίου του 2012 είναι όλα αυτά τα σκάφη τα οποία θα φεύγουν από τους κοινοτικούς λιμένες προκειμένου να λιεύσουν μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς απαραίτητα να αποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν τον ρόλο αυτό, θελούσια τουλάχιστον, να το δραματίσουν οργανώσεις παραγωγών. Δηλαδή αυτοί να έρθουν σε επαφή με τους αλείς και να θεσπίσουν ένα σύστημα βάσει του οποίου, για παράδειγμα, για μια συγκεκριμένη εβδομάδα θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό σκαφών με συγκεκριμένου αλληλεί που θα αλλιεύουν, την επόμενη εβδομάδα κάποιοι άλλοι. Κατά αυτόν τον τρόπο θα προσαρμόζονται καλύτερα στι ανάγκε τη αγορά. Γιατί διαφορετικά, όταν αλλιεύουν οι πάντε όλα τα σκάφη ανα πάσα στιγμή, καταλαβαίνετε ότι επηρεάζεται αρνητικά η ίδια αγορά στο τέλο. Ασκούνται πολύ αρνητικέ πιέσει στην αγορά. Θεωρώ λοιπόν ότι οργανώσει παραγωγών μπορούν να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και όσον αφορά τις ε, εισαγωγές, ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποτελούν αντικείμενο εισαγωγών όσον αφορά την κοινοτική μας αγορά. Νομίζω ότι εδώ, στον τομέα αυτό ακριβώς και για συγκεκριμένα είδη μπορούμε να πετύχουμε έναν καλύτερο συντονισμό με τις τρίτες χώρες από τις οποίες ε, εισάγουμε. Και θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε με αυτό και αυτή την ανάγκη την οποία θίγει ο Στρούαν Στίβενσον στην έκθεσή του όσον αφορά και τις περισσότερες πληροφορίες που θα πρέπει να έχουμε στα πλαίσια της αγοράς. Τώρα, τα περιφερειακά, ε, τα περιφερειακά συμβούλια λειτουργούν και συνεργάζονται προφανώς με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί κάπως το καθεστώ τους και να μπορούν να έχουν περαιτέρω αρμοδιότητες, όπως για παράδειγμα το να συλλέγουν περισσότερες πληροφορίες. Το έγγραφο αυτό είναι πάρα πολύ καλό, είναι εξαιρετικό και πραγματικά θέτει τις βάσεις για μια θετική μελλοντική εργασία όσον αφορά το ζήτημα αυτό, δηλαδή την κοινή οργάνωση αγορών στο τομέα της αλίας. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Στίβενσον για τη δουλειά που κάνατε, το έργο που επιτελέσατε ακόμα και για την επίσκεψη στην Ισπανία για να δείτε πώς έχουν τα πράγματα εκεί. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα επίσης να επισημάνω κάτι το οποίο πιστεύω ότι το είπαν και οι συνάδελφοι πιο πριν. Και αυτό είναι ότι σε αυτήν σε αυτή την πρόταση κανονισμού για την αναθεώρηση όσον αφορά την κοινή οργάνωση αγορών εξαφανίζεται απόλυτα η ανταλλαγή με τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική πολιτική. Ήταν ένα κεφάλαιο που βασιζόταν σε δασμολογικές προτιμήσεις ε, που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν καλά ε, δασμολογικά θέματα. Τώρα εξαφανίζεται αυτό. Τώρα, αυτό θα είναι γενική ε, αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Trade, εμπορίου. Όμως, θα διασφαλιστεί ένα σύστημα θα εξαφανιστεί ένα σύστημα το οποίο λειτουργήσε καλά, σχετικά καλά και το οποίο είχε εξισορροπήσει κάποια, κάποιους τομείς, για παράδειγμα της αλίας και της ε, επεξεργασίας. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι για το ότι δηλαδή είχαμε μια ε, κατάσταση που αν εξαφανιστεί αυτός ο ενδιάμεσος κρίκος μπορεί να έχουμε αρνητικέ επιπτώσεις. Μπορεί να διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε θα συνεχίσει να λειτουργεί ή να ζητηθεί από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να παρουσιάσει τις απόψεις ε, που έχει. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουμε στην κοινή οργάνωση αγοράς. Καθώς η Ευρώπη θέλουμε, είναι μια χώρα που όσον αφορά εισαγωγές εισάγει αλλιεύματα και έχει ανταλλαγές με τρίτες χώρες, αυτό αυτό είναι η ευρωπη θελουμε ειναι μια χωρα που οσον αφορα εισαγωγε εισαγει αλλιευματα και εχει ανταλλαγες με τριτες χωρες αυτο ειναι η λιδια λιθο τη μεταρρύθμισης και βρίσκεται ξαφνικά εκτό αρμοδιοτήτων τη επιτροπή μα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αποσαφινιστεί. Ποιο θα είναι ο αρμόδιο αν δεν είναι η Γενική Διεύθυνση που, ε, για την Αλία, να καλέσουμε τη Γενική Διεύθυνση για το Εμπόριο, να μα πει τι γίνεται με αυτού του μηχανισμού. Όσον αφορά, δεν θα κάνω λόγο ούτε για τα α, παράπλευρα αλλιεύματα που πρέπει να απορρίπτονται και να επιστρέφουν στη θάλασσα, ούτε για παρόμοια θέματα. Όσον αφορά εγώ, αυτό το θέμα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε τις διατομεακές, διακλαδικές ε, δράσεις ε, που ε, Όσον αφορά τις διατομεακές δράσεις, νομίζω είναι 4-5 συνολικά μανευρωπαϊκά. όμως όλος ο τομέας του, του τόνου, του ε, θήνου και για την επεξεργασία, μου φαίνεται ότι είναι οι πιο σωστές θέσεις ε, που μπορούν να εξεταστούν μέσω τέτοιων διατομεακών δράσεων. Είμαι υπέρ ε, εγώ αυτών των δράσεων όσον αφορά και τις ε, πολυεθνικές. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη δράση. Όσο υπάρχει μεγαλύτερη διατομιακή εμπλοκή, τόσο καλύτερη λειτουργία θα μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι σε ένα πολύ μικρό φάσμα θα μπορούμε να δράσουμε. Ενώ για τις διατομιακές και τις ε, υπερδια... Ε, πολυεθνικές δεν θα καλύπτονται οι πτυχές τους, τα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον έχουμε και ένα θέμα ετικετοποίησης και σημάτων. Γενικά η πρόταση για την κοινή οργάνωση αγοράς ε, και για τους μηχανισμούς παρέμβασης νομίζω ε, θετικά εξετάζεται. Είναι αρκετά καλή και σωστή η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλες οι παρεμβάσεις ε, σε σχέση με την ε, υποστήριξη αποθήκευσης για παράδειγμα όπως αναγνωρίζεται και από την Impact Assessment, τη μελέτη επιπτώσεων είναι θετικό αυτό το πλαίσιο και υποστηρίζω τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τις ετικέτες, ε, ετικετοποίηση υπάρχουν πρόοδοι σε σχέση με την πρόταση όμως δεν έχουν ληφθεί υπόψη πολλοί παράγοντες και κυρίως υπάρχει μια πτυχή για τα κατεψυγμένα και τα νόπα, είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση αυτών των αλλιευμάτων. Για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, όσον αφορά τους καταναλωτές, δεν είναι το ίδιο ένα σκάφος που ε, όσον αφορά την ημερομηνία αλίευσης, όσον έχει για παράδειγμα ε, τέτοιου είδους ε, υποχρεώσεις να καλύπτει τα αλλιεύματα με προηγούμενη ημερομηνία. Ενώ όταν έχουμε κατευσυγμένα όσον αφορά τον καταναλωτή η ημερομηνία μπορεί να δημιουργήσει κάποια σύγχυση για την πραγματική ημερομηνία σύλληψης, αλλίευσης των ε, αλλιευμάτων. Η ημερομηνία για παράδειγμα της εκφόρτωσης θα μπορούσε να εξεταστεί ως ε, λύση που θα μπορούσε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Η επισητιστική ασφάλεια είναι το θέμα. Ε, όχι ότι η ημερομηνία ή ε, μέσα σε μία περίοδο έξι μηνών όσον αφορά τα κατεψυγμένα θα δημιουργούσε πρόβλημα, αλλά μπορεί όλα αυτά να οδηγήσουν ε, σε αντιμετώπιση των κατεψυγμένων που δεν θα είναι ισοδίκαια. Υπάρχουν και προβλήματα τα οποία έχουν επισημανθεί από τον τομέα των αλλιέων και των, της, των κατεψυγμένων προϊόντων. Όμως όσον αφορά τα, την ετικετοποίηση πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα. Πρέπει να εξορθολογήσουμε όμως τις διεργασίες και να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές προτάσεις που έχει καταθέσει ο τομέας και που είναι πολλές φορές σωστές για την ετικετοποίηση. Πρέπει να πω ότι εδώ πάλι συμφωνώ με το impact assessment, με τις μελότητες επιπτώσεων, όπου λέει ότι διαβουλεύτηκαν με τον τομέα και διεκδικεί μεγαλύτερο δραστήριο ρόλο από τις αρχές και που θέλουν να υπάρχει ένα σαφέστερο πλαίσιο. Ένα σαφέστερο πλαίσιο το οποίο θα είναι πιο αποτελεσματικό. Σας διαβάζω τα όσα εμπεριέχονται στις συστάσεις αυτές υπάρχουν πάρα πολλές ιδιωτικές ετικέτες και όλες αυτές δημιουργούν πολλά προβλήματα και σύγχυση και δημιουργούν τεράστια σύγχυση όλες αυτές τις διαφορετικές ετικέτες ως αφορά τους καταναλωτές. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα, πρέπει να το πω. Και ζητήθηκε η οικοετικέτα, δηλαδή το οικολογικό σήμα και για τον Επίτροπο Φίσλερ που δεν ήταν, ας το πω έτσι, πυθύνιος και υποτακτικός, δημόσια αναγνώρισε εδώ ότι ένα από τα σφάλματά του ήταν ότι δεν μπόρεσε να επιβάλλει μία ενιαία ετικέτα, ένα ενιαίο σήμα στην Ευρώπη, λόγω των διαφορετικών πιέσεων που είχαν ασκηθεί από τις ιδιωτικές ετικέτες και ιδιωτικά σήματα. Πράγμα το οποίο παρακόλλησε και παρεμπόδισε το να υπάρξει συμφωνία για τα σήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε πια αυτό. Ε, το θέμα μιας ετικέτας, ένας, ενός ελάχιστου επίπεδου ευρωπαϊκής ετικέτας και ευρωπαϊκού σήματος που είναι απαραίτητο και πρέπει να γίνει. Θα ήταν η μόνη εγγύηση, τα μόνα ειχέγγυα για τους καταναλωτές έναντι, ας το πω έτσι, αυτού του χάους που έχει δημιουργηθεί ε, σήμερα στον τομέα αυτό. Και κάτι άλλο υπέρ της ε, αντιμετώπισης και καταπολέμησης της παράνομης και λαθρέας αλίας. Τα σήματα, οι ετικέτες θα έπρεπε να λάβουν υπόψη, να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα, να αναφέρεται το πιστοποιητικό αλίας που θα λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν είναι αλίευμα παράνομης ή λαθρέας αλίας. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε σχέση με τις νέες ετικέτες και τα νέα σήματα τα εισαγόμενα να διασφαλίζουν ότι δεν θα είναι ε, παράνομα αλλιεύματα και λαθρέα αλλιεύματα. Απαιτείται να γίνει αυτό σε ελάχιστη προϋπόθεση. Έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε καλύτερη ιχνηλασιμότητα και ανείχνευση σε σχέση με τον καταναλωτή να μπορεί να ξέρει πού ανάγεται αυτό το προϊόν, από πού προήλθε. Αυτά. Και τώρα από πλευρά τη Επιτροπή εσεί κύριε έχετε τον λόγο. Όχι, ο κύριο, τον κύριο Ραμπό είχαμε σημειώσει, αλλά εκεί όπου δεν υπάρχει καπετάνιο, ο, ο ναύτη, ο ναυτικό είναι το αφεντικό. Λοιπόν, we'll split the work between us. κύριο <laughs> Στίβενσον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και την καταπληκτική πληροφόρηση καθώ επίση και τα στοιχεία τα οποία μας εκδόβασαν και ευχαριστώ πραγματικά επίση και τα σχόλια τα οποία έχουν γίνει εδώ. Ακούσαμε πολλέ ερωτήσει και σας και επί τη ουσία και θέματα από τη πολιτική. Θα ήθελα να αφαιράσω, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Λαμπό, θα ήθελα να πω το εξή. Αναφερθήκατε στην έλλειψη έλλειψη ε, πολιτικής σε αυτή τη, τον Δεν θα θέλαμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα κείμενο το οποίο απομονώνει το εμπόριο και μόνο. Αυτή είναι η νομική δομή του όλου κειμένου και πιστεύω πως είναι νομοθετικό κείμενο το οποίο αυτή τη στιγμή να μπορεί να καλύψει όλα εκείνα τα προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορή, μη πω καλά συνθήκας και με τεχνική πλευρά θα λέγαμε ότι είναι, είναι ένας αυτοματισμός ο οποίος τίθεται αυτή τη στιγμή των ποσοστώσεων μέσα στον κανονισμό. Δεν θα ήθελα να περάσω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται από δύο γενικές διευθύνσεις και προσπαθήσαμε να ενοποιήσουμε αυτούς τους κανονισμούς και αυτή είναι η εργασία που έχει γίνει προς στιγμή. Επίσης θα ήθελα να πω πως αυτό είναι ένα νομοθετικό κείμενο οποία αναγγέλει που είχε αναγγελθεί στην αναγγελία όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και είχε λεχθεί αυτό το. Και κατά αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω στον Χριστιανό Λομπό να συνεχίσει με τα κατηδίαν ερωτήματα τα οποία τέθηκαν πιθανότητας αυτού. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν και με βάση το κείμενο του κ. Στίβεντο το καταπληκτική έκθεση. Πιστεύω πως υπογραμμίσατε όλη την ανάγκη ότι η πρόταση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επιτρέψει να καλύψει, αν θέλετε, όλες τις περιπτώσεις και τις περιπτωσιολογίες και αυτό θα είναι μια νέα δυναμική η οποία θα απορροφηθεί ανάλογα με την εισαγωγή αυτή τη κοινή ε, πολιτική πολιτικής. Επίσης το ερώτημα κύριε Στέβεν, κατά πόσο οι, οργανώσεις των παραγωγών έχουν ένα ρόλο να παίξουν όσον αφορά τι εκχωρήσει που γίνεται. Κανονικά θα έλεγα ότι ενωμένοι νικάμε. Και αν δεν συμβαίνει αυτό πάντοτε, θα πρέπει να πιστέψουμε ότι αν υπάρξει μια αμοιβαιότητα στα πλαίσια μιας επαγγελματικής οργάνωσης, παραγωγών προκειμένου, καθώς επίσης και η συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων θα διευκολύνει την συντήρηση ή την αύξηση των διαφόρων, της δύναμης των διαφόρων παραγωγών. Τώρα, όσον αφορά το πρόβλημα της εγκατάστασης των παραγωγικών ομάδων, θα πρέπει να σας πω, έχουμε 214 στο σύνολο. Εσείς δώσατε ορισμένους αριθμούς προηγουμένως για την διδακολία, και την αλληλεία. Σε ορισμένε χώρε, αυτέ οι οργανώσει παραγωγού εκπροσωπούν το 80% των ε, αλληλευμάτων που φτάνουν στην αποθήκη. Είναι άνισα τα πράγματα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω, διότι οι οργανώσει παραγωγών δεν είχαν μέχρι στιγμή ένα ρόλο καθοριστικό για την ανάπτυξή του. Η ιδέα τώρα λοιπόν με αυτή τη μεταρρύθμιση που έχουμε αναχείρα είναι να μπορέσει να υπάρξει μια επαναδιατύπωση καθώς επίσης και δίνοντας μέτρα συμπληρωματικά για να παίξουν αυτό το ρόλο που δεν έπαιζαν μέχρι τούδε θα ενδεχομένως αναπτυχθούν στα κράτη-μέλη ε, και ιδιαίτερα σε εκείνες χώρες οι οποίες δεν ήταν και πιο θερμές. Επίσης ο κ. Στίβενσον είπε το εξή και αυτό απαιτείται και άλλο παρεμβάσιο που έγινε παρεμπιπτόντων, κατά πόσο η αυτή τη στιγμή, η Κομισιόν μάλλον, απέφυγε να μιλήσει για τη συγχώνευση και την αναδιάρθρωση τόσο για τους παραγωγούς όσο και στα κράτη-μέλη, όσο και τις, τους, ε, των κυβερνών των εκείνων οργανισμών, γιατί δεν θα πούμε εμεί πώ θα γίνει ένα αναδιάρθρωση και ένα αναδιοργάνωση. Διότι η πρόταση τη Κομισιόν αυτή τη στιγμή, σαν σκοπό, έχει να δοθεί μια νέα ζωή σε αυτέ τι ε, συνεταιρισμού οργανώσει που υπάρχουν, να γίνει δηλαδή με έναν τρόπο πολύ πιο ομαδικό μεταξύ των διαφόρων χωρών και να υπάρχει μέτρα. μέτρα. Αυτό το νέο μέτρο λοιπόν θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία. Τώρα όσον αφορά τα απόβλητα, τις παρα... πλε... παράπλευρες αλλιεύσεις, ξέρετε, ο αποτέλεσμα είναι διπλό. Καταρχήν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναλάβουν οι οργανώσεις παραγωγής τη ροή αυτών. Όχι, δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι σε αυτή την αποστολή που δίδει στις οργανώσεις των παραγωγών είναι να γίνει μια τέτοια αναδόμηση ώστε να υπάρξει μια βιώσιμη αλλιεύση. Να μειωθούν αυτές οι παράπλευρες αλλίες, αυτός είναι ο σκοπός και αυτή είναι η αποστολή της, ούτως ώστε να υπάρξει μια καλύτερη ροή, ότι θα πρέπει να γίνεται μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, ετήσια βεβαίω, και τα πράγματα πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα εξαφανίσουν τα υπάρχοντα οι, ε, οι προτάσεις αυτές θα μειώσουν τα υπάρχοντα προβλήματα. Τώρα όσον αφορά το θέμα της διανομής στους διαφόρους παραγωγούς, το σύστημα είναι σε θελούσια βάση. Δεν υπάρχει τίποτα το υποχρεωτικό, είναι ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει ήδη και το οποίο διατηρείται. Τόσο αφορά την διανομή που γίνεται για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η τις οργανωσεις υπάρχει, δεν θα θέλαμε να γίνει αυτή τη στιγμή ένα νέο εργαλείο, αλλά λέμε εάν υπάρξει ανάγκη, κάλλιστα θα μπορούσαν να επιτραπούν να, υπάρξει, να υπάρχει τέτοιου είδους ροή των παρααλλιευμάτων. Αναφερθήκατε προηγουμένω και στέβες όσον αφορά στον εξυγχρονισμό τη αλληλείας, τη δυνατότητε που υπάρχουν προσφυγών κλπ. Σα υπενθυμίζω λοιπόν πώ. Καταρχήν είναι εργαλεία τα οποία είναι ευανάγνωστα και υπάρχουν και παρεμένω όπως έχουν μέσα στην πρόταση που έχουμε αυτή τη στιγμή και θεωρούμε πως οι οργανώσεις παραγωγών ή οποιοδήποτε άλλος έχουν σαν αποστολή να διευκολύνουν ε. Όσον αφορά το σύστημα ενισχύσεων για την αποθήκευση, πολλοί πήρανε το λόγο για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο μηχανισμός. Συμφωνούμε όλοι ως προς αυτό αλλά θα πρέπει να καταργηθούν οι δημόσιες δαπάνες όσον αφορά την καταστροφή των ελευμάτων. Αυτό αποτελεί πολύ θετικό βήμα. Ο μηχανισμός δεν γίνεται κατανοητός αν διαβάσουμε απλώς τον κανονισμό κοινή οργάνωσης αγοράς. Θα πρέπει να δούμε και τον κανονισμό μάλλον και την ε, πρόταση η οποία συνοδεύει το σύστημα αυτό όσον αφορά την χρηματοδότησή του για το οικολογικό σήμα τώρα. Ξέρετε ότι η ε, κυρία Φράγκα στο παρελθόν ε, υπήρχαν πολλοί οι οποίοι δεν θέλαν να ακολουθήσουμε το δρόμο αυτό του οικολογικού σήματος. Δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Να πω μόνο ότι δίστανται οι απόψεις καλύπτονται όλες οι διαφορετικές τοποθετήσεις όσον αφορά το σύστημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια στην πρότασή μας όσον αφορά το ζήτημα της ετικετοθεσίας. Και οι τρεις στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να επανεληφθούν εδώ πέρα μια ακόμη φορά. Πρώτον, πρώτος στόχος, να ενημερώσουμε τον καταναλωτή, να διευκολύνουμε την επιλογή του καταναλωτή όταν βρίσκεται ενώπιον των διαθέσιμων προϊόντων. Δεύτερον, να επιτρέψουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα στα προϊόντα και κύριε Μιλενάρα, η ημερομηνία αλίευσης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης, αποτελεί θετική διακριτική μεταχείριση, αν θέλετε, για συγκεκριμένα προϊόντα, για κάποια νοπά προϊόντα και ουσιαστικά διακρίνει θετικά υπέρ των νοπών ελευτικών προϊόντων σε σχέση με τα κατεψυγμένα αυτά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και που παρουσιάζονται σαν να ήταν φρέσκα στο ηχθειοπολείο. Ένα άλλο στοιχείο θετικής διακριτικής μεταχείρισης είναι το ακόλουθο. Όλοι εδώ πέρα αλλά και αλλού είμαστε υπέρ ενός συστήματος που θα είναι υπέρ της αλίας μικρούς κλίμακας της βιοτεχνικής αλίας. Αν θέλετε να προωθήσουμε πραγματικά τους μικρούς παραγωγούς, μπορούμε να τους βοηθήσουμε χρησιμοποιώντας την ημερομηνία αλίευσης. Θα καταφέρουμε πάλι να διαφοροποιήσουμε το προϊόν αυτό, το οποίο έχει περάσει 24 ώρες μόνο στο σκάφος, σε σχέση με αυτό που έχει περάσει 15 μέρες πάνω στο σκάφος. Ενδεχομένως να ευνοούμε κάποιους και άλλους να τους λιγότερο, αλλά έπρεπε να πάρουμε την απόφαση αυτή. Επίση, θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένε ενδείξει σε συγκεκριμένα προϊόντα όπω οι κονσέρβε. Στο παρελθόν αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα. Αν καταφέρουμε να ενημερώνουμε τον καταναλωτή για την ζώνη αλίευση, τότε μπορεί ο καταναλωτή να γνωρίζει ποια είναι η προέλευση του προϊόντο. Η προέλευση ε, του ε, προϊόντος είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, Νομίζω ότι ο συνάδελφός μου σας απάντησε ήδη για το ζήτημα αυτό, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Σας ε, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας όσον αφορά την πρόταση αυτή για την συλλογή περισσότερων πληροφοριών. Μέχρι ε, το επόμενο έτος ε, το παρατηρητήριο αυτό το οποίο αποτελεί ουσιαστικά πρόταση της δικής σας Επιτροπής. Είναι ένα σχέδιο το οποίο θα ξεκινήσει και στα τέλη του 2012 ελπίζω ότι θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τα πρώτα συμπεράσματα του παρατηρητηρίου αυτού. Όσον αφορά τώρα την αλία και την καλλιέργεια, Νομίζω ότι για πρώτη φορά στα πλαίσια των κοινών οργανώσεων αγορών καταφέρνουμε να διακρίνουμε και να αναγνωρίσουμε και τους δύο τομεί επαγγελματιών, τους αλείς δηλαδή και τους υδατοκαλλιεργητέ. Και μπορούμε πραγματικά να κάνουμε μια σαφή διάκριση ανάμεσα στι δύο αυτέ κατηγορίε επαγγελματιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το υπογραμμίζω. Κύριε Καντέκα, σας ευχαριστώ για τη δική σας την υποστήριξη. Να προσθέσω μόνο κάτι, να συμπληρώσω αν θέλετε την πρότασή σας όσον αφορά την ε, τιμή ε, εκκίνησης καθώς επίσης και το μηχανισμό βοήθειας υποστήριξης όσον αφορά την αποθήκευση. Σε σχέση με το νέο αυτό χρηματοδοτικό μέσο, λοιπόν, τα ποσά τα οποία παρατίθενται, δηλαδή 45 εκατομμύρια ευρώ για τα πέντε πρώτα χρόνια υπέρ της, ε, του μηχανισμού αποθήκευσης, αντιστοιχούν ακριβώς στο, στην υφιστάμενη κατάσταση, ως σημείο κίνησης τουλάχιστον. Το σύστημα είναι απόλυτα αναλογικό. Σε καμία περίπτωση θα υπάρξει μια υπερβολική δημόσια χρηματοδότηση όσον αφορά το σύστημα υποστήριξης αποθήκευσης. Υπάρχει μάλιστα και ένα σύστημα το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα ανώτατα όρια τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Επομένω, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο, ούτε θα έχουμε σημαντική αύξηση τη δημόσια δαπάνη για το σύστημα αυτό, ούτε θα έχουμε αύξηση των ε, αλλιευμάτων αυτών που καταλήγουν στα ευρωπαϊκά ψυγεία, να το θέσω έτσι ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες αδυναμίες όσον αφορά την υποδομή, σε καμία περίπτωση θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε ψυγεία σε όλους τους λιμένες. Καθησυχάζω προς αυτό. Και κάτι ακόμα, συγχωρήστε με αν μένω τόσο πολύ στο σημείο αυτό. Αν η βοήθεια που προβλέπετε είναι ε, αντίστροφα ανάλογη για το σύστημα αυτό της αποθήκευσης, αυτό προβλέπεται ακριβώς επειδή ουσιαστικά θέλουμε να εκμηδενήσουμε κάθε παρέμβαση στην αγορά. Θέλουμε να διοργανώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την ελευτική δραστηριότητα ώστε να ανταποκρίνεται, να συνάδει με τις ανάγκες της αγοράς. Κάτι ακόμα όσον αφορά την παράνομη λαθρέα αναρχιαλία, η κυρία Φράγκα. Ένα προϊόν το οποίο εισάγεται και το οποίο δεν συνοδεύεται από πιστοποιητικό δεν μπορεί να εισέλθει στο, στην κοινοτική επικράτεια. Επομένως, δεν τίθεται καν το ζήτημα του ζήματος, γιατί εφόσον διατεθεί στην αγορά πρόκειται για, καθαρά, για, για καθαρή απάτη. Κάθε προϊόν το οποίο εισάγεται στο κοινοτικό έδαφος θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά. Και αυτό γίνεται με όλα τα ψάρια τα οποία πολλούνται. Πρόκειται για νόμιμη αλία αναγκαστικά. Γι' αυτό το λόγο δεν προβλέπεται ένα πιστοποιητικό σε σχέση με την παράνομη και ελαφραία αλία. Πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, πως απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που θέτησα. Μάλιστα. Θα ήθελα να επανέλθω και να εμείνω, να επιμείνω ποια είναι η νομική βάση αυτού του κανονισμού. Αποκινούμε την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για τις συναλλαγές με τρίτες χώρες. Είναι εμπορική πολιτική ή αλλιευτική πολιτική η νομική βάση. Ποια νομική βάση υπάρχει. Άρθρο 31. Δεν είναι όσον αφορά τους φόρους, αλλά είναι το άρθρο 31 Ε, eh, Μάλιστα, ο κύριος Στίβενσον, Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν και με σημειώσεις ε, που έγιναν πλήρης και ε, άκουσα κύριε Λεβίν ότι κερδίσαμε και κάποια, κάποιες πιστώσεις, κάποιες ας το πω έτσι μεταφραστικές ας το πω έτσι άρετες για την έκθεσή μου, επειδή υπήρξαν και μεταφραστικά θετικά στοιχεία και σε σχέση με την έκθεση που είχε διανεμηθεί. Χρησιμοποίησα όλα αυτά τα στοιχεία και νομίζω τώρα ότι έχουμε φτάσει στο ε, αρχικό επίπεδο. Το συγκεκριμένο ακριβώς σημείο το οποίο θίξατε στην παρέμβασή σας για το με ποιους ε, υπήρξε επαφή. Ακούσατε, όταν δόθηκε αυτή η έκθεση αποφάσισα να πάω στην Γαλλικία, της Ισπανίας, διότι το ίμιση των διευθύνσεων και των οργανισμών αυτών βρίσκονται στην ε, Ισπανία σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών αλληλείας ε, και υδατοκαλλιέργειας. 110 βρίσκονται στη Γαλλικία και μίλησα και με μια ολόκληρη σειρά υπουργών. Είχα και ένα εργαστήριο, workshop, όπου με όλους τους κοιόδης εισηγητές ε, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την οικονομική πτυχή της αλίας και οικονομολογική, ας το πω έτσι, συνεισφορά, συνάντησα και εκπροσώπους από την Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Αγγλία, Σκοτία και με μια σειρά πλοιάρχων και για την επεξεργασία αρμόδιου συνάντησα πήγα σε πολύ διαφορετικές αγορές ηλεκτρονικές αγορές και τις μεγαλύτερες αγορές όπου επιφυλάσσονται να κάνουν χρήση τέτοιου είδους ε, προοπτικών. Μίλησα με μια ολόκληρη σειρά ΜΚΟ και εμπλεκόμενος. Και είχα μια ολόκληρη σειρά συναντήσεων και επισκέψεων που απομένουν ακόμα. Τον Ιανουάριο θα επισκεφθώ την Ολλανδία και θα συναντήσω εκεί εκπροσώπους των αλλιέων και κάποιοι Πολωνοί επίσης αλληλείς ε, με τις συναντήσεις που προβλέπονται θα εισακουστούν. Και τώρα με όλες αυτές τις πολυσχηδείς δραστηριότητες ε, είμαι πρόθυμος να συναντήσω οποιονδήποτε θέλει να έρθει και να μου πει οτιδήποτε. Πολλά από αυτά λοιπόν για την αναθεώρηση του εγγράφου εργασίας και ίσως τον Ιανουάριο θα πρέπει να συνέρθουμε με τους σκιώδεις συζητητές και να δούμε αν μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο μακριά με το θέμα της έκθεσης. Και επίσης ε, πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μεγάλη εμπλοκή με τη δική σας έκθεση, κυρία, διότι αυτά τα οποία εσείς εξετάζετε έχουν επιπτώσεις και σε αυτά τα οποία εξετάζω εγώ. Ο συντονισμός μεταξύ των δύο, των δύο μας θα ήταν θετικός. Ευχαριστώ λοιπόν για όλα τα σχόλιά σας. Bueno, pues, πολύ καλά λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Στίβενσον. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Ντεπίπερ και ολοκληρώθηκε η εξέταση εδώ του σημείου 7 του σημείου 7 της σημερισίας διάταξης. Θα συνεχίσουμε με τη συζήτηση του θέματος βέβαια. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα στην ημερησία διάταξη για απόψε. Θα λήξει η συνεδρίαση. Υπενθυμίζω σε όλους σας όμως πιο πριν ότι στις 6.30 έχουμε το κόκτέιλ για τα Χριστούγεννα. Θα έρθει η Επίτροπος Δαμανάκη επίσης. Είναι αυτονόητο, είναι φυσικό ότι είσαστε προσκεκλημένοι όλοι σας και οι διερμηνείς και όλοι οι υπάλληλοι σε αυτό το κόκτελ στις 6.30 στο μπαρ των Ευρωβουλευτών, στο εστιατόριο των Ευρωβουλευτών. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο. Ελπίζω να έρθετε. Αύριο στις 9 θα έχουμε το workshop, το εργαστήριο με τα ε, θαλάσσια οικοσυστήματα. Λίγη συνεδρίασή μας. Γεια σας.